Ladies and Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Να αρχίσουμε με τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και σας τους συναδέλφους και τους βοηθούς και τους προσκεκλημένους. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο ζωντανά. Και η προτεραιότητα και το γλωσσικό καθεστώς δίνεται στα τακτικά μέλη της ε, Επιτροπής μας. Η μερίσια διάταξη για σήμερα έχει διανεμηθεί. Και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, υποθέτω ότι εγκρίνεται. Θα ήθελα να εγκρίνουμε τα πρακτικά των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων. 28 Μαΐου, 16 και 17 Ιουνίου. Αν θέλετε να κάνετε σχόλια, παρατηρήσεις ε, ή να εκφράσετε επιφυλάξεις, ε, παρακαλώ να το κάνετε μέχρι το πέρας της ε, σημερινής συνεδρίασης. Να περάσουμε τώρα στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή τη ΕΕΔ, τον κύριο Βοπόφσκι, Έχετε πολλές φορές παρευρεθεί σε συνεδριάσεις μας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι. Θα ήθελα να μας πείτε ορισμένα πράγματα για τις προοπτικές, για την ΚΠΑ, κατόπιν ε, της ε, πρόσφατης Ευρωπαϊκής Συνόδου. Θα θέλαμε ο πρέσβης Ποπόφσκι να μας ε, συνοψίσει τα συμπεράσματα της ε, Συνόδου και να μας ενημερώσει για ε, τις διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ποπόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι και πάλι εδώ Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε ασχοληθεί σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, με την ε, ΚΠΑ. Ε, τελικά αυτό δεν έγινε για πολλούς λόγους, θα επανέλθω σε αυτό. Πάντως ανανεώσαμε τη δέσμευσή μας για να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, στο πλαίσιο ενός περιβάλλον που, ενός περιβάλλοντος που επιδεινώνεται από από απόψεως ασφαλείας. Εμείς ζητήσαμε από την ύπατη εκπρόσωπο να αναπτύξει μια παγκόσμια στρατηγική μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Πράγματι ε, παρουσιάστηκε το πρώτο τμήμα μιας στρατηγικής αυτής, η αξιολόγηση του ε, περιβάλλοντος ασφαλείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το Συμβούλιο θα υπάρξει βέβαια και μια πολύ μεγάλη διαδικασία με δύο σκέλη διαβουλεύσεων, ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως και με ε, think tanks και ε, ακαδημαϊκούς, μπορεί να πάρει κάποιους μήνες και θα υπάρξει και ένα νέο πλαίσιο το οποίο ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Εκτός από την ανανέωση της δέσμευσης ε, για την ΚΠΑ, την ε, ε, ανάπτυξη υποδομών που χρειάζεται η Ευρώπη και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, η αρχική ιδέα ήταν να ασχοληθούμε περισσότερο με την ασφάλεια και την άμενη άμυνα, όμως επειδή υπήρξε αυτή η τεράστια κρίση με την Ελλάδα και το μεταναστευτικό κύμα. Ε, δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε όσο θέλαμε, αλλά έγινε μία συζήτηση. Καταρχάς, ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ε, έγινε ανταλλαγή απόψεων με τους ηγέτες. Αυτό έγινε στις 26 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Και επίσης οι ηγέτες επικεντρώθηκαν σε μερικά συγκεκριμένα ζητήματα στο σχέδιο συμπερασμάτων. Υπήρξε μια ανταλλαγή απόψε, όχι τόσο ζωηρή όσο το Δεκέμβριο του 2013, αλλά έγινε και τα συμπεράσματα μπορεί να ήταν πάρα πολύ σύντομα, αλλά υπήρχε αυτή η γενική τάση, ε, υπάρχει αυτή η γενική τάση να είναι συνοπτικά τα συμπεράσματα πλέον. Έχουν παρόλα αυτά συμπεριλάβει τα βασικά μηνύματα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, επανεπιβεβαίωση των συμπερασμάτων ε, των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης το Μάιο, δεν... Ε, Χρειάστηκε, δεν χρειάζεται να πω σε πολλέ λεπτομέρειε, το είχαμε ε, αναφέρει την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ. Υπάρχει ένα κατάλογο στρατηγικών, στρατηγικών στόχων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, παγκόσμια στρατηγική, όπω είπα και προηγουμένω. Υπάρχει μια υπόσχεση για περισσότερες επενδύσεις ε, στην άμυνα. Αναγνώριση ότι η Ευρώπη ε, χρειάζονται περισσότερες δαπάνες με καλύτερο τρόπο χωρίς να αλλάξουμε ε, τα ονομαστικά ποσά του ΝΑΤΟ γιατί αυτό είναι κάτι επειδή υπάρχουν κάποια μέλη της Ένωσης που είναι μέλη και της Συμμαχίας, προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις αμυντικές δαπάνες της Ένωσης με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Υπήρχε μια σημαντική συζήτηση για την κινητοποίηση ε, ενωσιακών κονδυλίων, για την ενίσχυση της ε, αμυντικής στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη μνήμα για το θέμα αυτό, ώστε να υπάρξει μια προπαρασκευαστική δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία ενός προγράμματος προαγγέλου για την έρευνα και την ανάπτυξη και για την άμυνα υπάρχουν προσωπικότητες που καθοδηγούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση, τον προϋπολογισμό μεταξύ των οποίων είναι και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και της βιομηχανίας ε, και των κρατών μελών αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Αν όλα πάνε καλά, αυτή η προπαρασκευαστική, δράση θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή το 2017 και θα μπορούσε τότε να μετατραπεί σε μια ε, γραμμή προϋπολογισμού συγκεκριμένα για την άμυνα υπό το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στους Υπουργούς Άμυνας το Νοέμβριο. Επίσης ε, γίνεται πολλή δουλειά για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και και για την ασφάλεια του ε, ανεφοδιασμού στον αμυντικό τομέα. Οι ηγέτες αναγνώρισαν ε, τη μεγάλη απειλή ε, λόγω των υβριδικών τακτικών του υβριδικού πολέμου. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κατέληξαν σε μία στρατηγική για το πώς να το αντιμετωπίσουν. Ε, υπάρχει λοιπόν καθήκον το οποίο επιφορτίζει την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, για να υπάρξει στατιστική στρατηγική για το θέμα αυτό μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Καταρχά, το θέμα του κατά πόσο ε, είμαστε ευαισθητοποιημένοι για την κατάσταση αυτή, ότι υπάρχει δηλαδή απειλή γύρω από την Ευρώπη στην Ευρώπη και πώ μπορούμε να αυξήσουμε την αντοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιου είδου ε, καταστάσει. Πώ να προστατεύσουμε, για παράδειγμα, κριτικέ κρίσιμε υποδομέ, ε, πώ να αντιμετωπίσουμε επιθετική προπαγάνδα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Πρέπει να υπάρξει πλαίσιο που θα αναπτυχθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχουμε καθυστερήσει σε κάποιου τομεί, και επίσης ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνα θα συμμετέχει και εκείνο. Είναι ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος ε, και για το ΝΑΤΟ και έχουμε ήδη ανταλλαγές απόψεων χρήσιμες με τους συναδέλφους ε, από το Διεθνές Προσωπικό του ΝΑΤΟ. Υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης ε, για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοφόρο, στον κυβερνοχώρο, για θέματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης υποδομών κλπ. Εκ νέου λοιπόν αναφέραμε τη δέσμευσή μας ε, για τη σημασία της συνεργασίας. Ε, η συνεργασία σημαίνει προφανώς με, με άλλους οργανισμούς, ανέφερθηκα στην Αφρικανική Ένωση, στο ΝΑΤΟ και με χώρες εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ. Και αυτό είναι μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία ε, η οποία τονίστηκε από τους ηγέτες. Είναι μία πρωτοβουλία που την αποκαλούσαμε εκπαίδευση και εξοπλισμό, train and equip. Ε, είναι σημαντική στον τομέα της ε, ανάπτυξης της ασφάλειας ε, και είναι μια ιδέα που την παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο, βασικό στόχος είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους, ε, στις χώρες εταίρους να αναλάβουν μόνοι τους την ασφάλειά τους. Μαλή, Σομαλία, ε, Αφρικανική Ένωση, είναι πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο να μπορεί να συμβεί. Δεν μιλάμε μόνο για την ε, Αφρική βέβαια, δεν θέλουμε η πρωτοβουλία αυτή να εξαντλείται στην Αφρική, θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες εταίρους σε όλο τον κόσμο. Οπότε τώρα εξετάζουμε Καταρχάς, επακριβώς τα διάφορα ε, προγράμματα στα ε, διάφορα κράτη, τι κάνουν τα κράτη-μέλη, τι κάνουμε εμείς με τις αποστολές μας και τις επιχειρήσεις μας, προσπαθούμε να μάθουμε από πιλωτικές περιπτώσεις όπως το Μαλί και η Σομαλία και όταν υπάρχει ανάγκη προσπαθούμε να υπάρξει ένα μέσο χρηματοδοτικό ειδικό το οποίο βοηθά την ανάπτυξη ε, υποδομών αμυντικών ε, και ασφαλείας ε, στις χώρες μέλη. Είχαμε ήδη συζητήσεις με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευκαιρία θα είναι η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του οικονομικού πλαισίου, υποθέτω κατά τα, κατά τα μέσα προς τέλη του επόμενου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα αποφασίσει αυτό. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι υπάρχει και πολιτική όθηση για τη συνέχιση της ε, δουλειάς για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αναφέρθηκα στο προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα και την ανάπτυξη ή για την εκπαίδευση και εξοπλισμό. Ε, πρέπει όμως να ε, καρποφορήσουν όλα αυτά που είπαμε το 2013. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παραμείνει ε, δεσμευμένο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά αυτή ήταν ε, η πρόθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραμείνει η δέσμευση ε, να επιτρέψει ε, στα κράτη-μέλη να επανέλθουν στη συζήτηση για την άμυνα και την ασφάλεια, για την αναθεώρηση της προόδου και για να υπάρξει και περαιτέρω καθοδήγηση. Θα γίνει κάτι τέτοιο τον Ιούνιο του 2016 για να υπάρξει συζήτηση και ελπίζουμε να ε, εγκρίνουμε και την νέα στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πλήρη παρουσίαση σήμερα το πρωί. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές, τις οποίες καλείστε να απαντήσετε. Τα μέλη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να υποβάλουν τώρα ερωτήσεις. Θα αρχίσουμε με τους συντονιστές που είναι παρόντες Σλέζινγκ και μετά η κυρία Βαλέρ. Ευχαριστώ. Μιλάω γερμανικά, με ακούτε. Κάποιες ερωτήσεις για αυτά που είπατε. Είπατε ότι δώσατε εντολή στην κυρία Μογκερίνη να χαράξει μια παγκόσμια στρατηγική για την ασφάλεια και άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είδους είναι αυτό το έγγραφο που περιμένετε. Πρόκειται για μια νέα ε, στρατηγική ασφάλειας της ε, Ευρωπαϊκής Υπήρου. Υπήρχαν και παλιότερα προσπάθειες να χαραχτεί μια τέτοια πολιτική και ε, ως γνωστόν απέτυχαν οι προσπάθειες αυτές. Οπότε, εσείς γιατί πιστεύετε ότι αυτή η νέα προσπάθεια έχει καλύτερες πιθανότητες να πετύχει ή σε τι διαφέρει αυτή η νέα προσπάθεια από τις παλαιότερες. Επίσης, είπατε ότι ζητούμενο είναι να υπάρχει μια συστηματική ε, συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η οποία ε, θα πρέπει να χρηματοδοτείται και με ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να διαθέτει και ορισμένες βασικές, σημαντικές ικανότητες, δυνατότητες. Σε ποιες ακριβώς δυνατότητες αναφέρεστε και τι ύψους χρηματοδότηση αναμένεται. Και στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι η κατάλληλη ε, χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών ε, εργασιών θα πρέπει να διασφαλιστεί για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Για τι, είδους, τι ύψους ποσά μιλάμε. Αυτές οι, οι προπαρασκευαστικές εργασίες ε, εντάσσεται στην γραμμή ε, του προϋπολογισμού για τους εξοπλισμούς. Εσείς ποιο είναι το ποσό που πιστεύετε ότι θα μπορούσε ή θα έπρεπε να χρηματοδοτεί ε, αυτές τις δραστηριότητες. Uh, all the best. Σας ε, εύχομαι καταρχήν να σας συγχαρώ για τη θέση σας και έχετε το λόγο κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ θα μιλήσω σου ειδικά σήμερα το πρωί, άρα σας παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά. Θα ήθελα να αναφερθώ στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του 2013, γιατί στα νέα συμπεράσματα γίνεται μνήα στη συνάντηση αυτή του Δεκεμβρίου του 2013 και θυμάμαι ότι όταν διάβασα εκείνα τα συμπεράσματα ε, μιλήσαμε για μια ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όπλων και μιλήσαμε και για ε, μια εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση γιατί μιλάμε και για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πολιτική άμυνας καθαρά των ευρωπαϊκών κρατών και όχι για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Άρα η βιομηχανία ευρωπαϊκών εξοπλισμών ή όπλων είναι κατακαιρματισμένη και δεν συνεργαζόμαστε, δεν υπάρχει συνεργατική πολιτική. Άρα εξαρτόμαστε από τις εξαγωγές μας. Ξέρω ότι θα το συζητήσουμε αργότερα σήμερα το πρωί. Γνωμοδοτήσαμε στο Κοινοβούλιο σε μια έκθεση της Αναγκόμες, η οποία είπε ότι δεν πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων, απλώς θα πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα οι χώρες μεταξύ τους. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γνωρίζουμε ότι δεν θα προωθήσουμε την άμυνά μας προωθώντας τη βιομηχανία όπλων, αλλά θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με μια ποιοτική εργασία. Και ήθελα να ρωτήσω πώς προσεγγίζεται το θέμα της ποιότητας μέσα στα πλαίσια της αμυντικής μας ικανότητας, γιατί δεν μιλάμε για περισσότερα όπλα, αλλά για καλύτερη χρήση των υπαρχόντων. Αυτό το 2% του ΑΕΠ, αυτό το στόχο τον ακούμε συνεχώς καλείται τους πάντες να αυξήσουν τον προϋπολογισμό άμυνας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαθέτουν και καλύτερη άμυνα. Άρα μας ενδιαφέρει η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Θίξαμε και δημοσιονομικά ζητήματα. Εδώ μας ενδιαφέρει η έρευνα, η πτυχή της έρευνας Επίσης, περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για την έρευνα, για την άμυνα. Αυτό όμως σημαίνει ότι παίρνουμε χρήματα από την πολιτική άμυνα. Ο κύριος Γιούρεκ, ο Μάρεκ Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποβάλω ένα καθαρά πρακτικό, πρακτική υφής ερώτημα. Στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έγινε μια ανακοίνωση ότι θα αναλάβουμε στρατιωτική δράση κατά των λαθρεμπόρων στη Βόρεια Αφρική. Αλλά δυστυχώς ε, τίποτα δεν έγινε γιατί δεν υπάρχει εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη. Έγινε κάτι έκτοτε για να λάβουμε την εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη και θα σταματήσουμε αυτή τη δραστηριότητα στη Βόρειο Αφρική. Το λαθρεμπόριο και την δουλεμπορία δηλαδή. Το δουλεμπόριο τι θα γίνει τα ερχόμενα χρόνια στην νότια, στις νότιες όχθες μας της Μεσογείου. Οι δηλώσεις του πρώτου τελευταίου συμβουλίου είναι ε, νεκρά λόγια είναι λόγια επιχάρτου ή ουσίας. Ο κύριος ε, Κρέντσα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, πρεσβευτή Ποπόφσκι, ο οποίος ε, σήμερα το πρωί μας μίλησε για την κατάσταση στην πολιτική άμυνας. Πιστεύω, σε σχέση με τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας, που είναι οικονομική υφής και εδώ αναφέρομαι στην Ελλάδα, οι προκλήσεις αφορούν τη μετανάστευση η οποία διονγκούται. Μιλώ για την παράνομη μετανάστευση. Ξέρετε ότι στην Ιταλία έχουμε πληγεί πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες. Και σε σχέση με την πρόκληση της τρομοκρατίας πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη δηλαδή να έχουμε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη εξωτερική πολιτική που θα πρέπει να αναθέσουμε στην ύπατη εκπρόσωπό μας, δηλαδή η δύναμη για μια πραγματική εξωτερική πολιτική. Χαίρομαι γιατί βρίσκομαι εδώ από το 2004 και ξέρω ότι και βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις στην πολιτική άμυνας θα πρέπει να την προωθήσουμε σε σχέση με τις προκλήσεις που προανέφερα. Είδατε τα έγγραφα του 2013, 14 και 15. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις. Και σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λούζιγκερ, σε σχέση με το θέμα των πόρων. Τι κάνουμε ακριβώς έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τις ε, πολιτικές αυτές ενίσχυσης της ε, πολιτικής έρευνας, της έρευνάς μας, της ευρωπαϊκής έρευνας. Εγώ είμαι ειρηνιστής, αλλά ενώπιον ορισμένων φαινομένων μπορούμε να πούμε ότι αν δεν διαθέτουμε τα μέσα δεν θα μπορέσουμε, τα κατάλληλα μέσα δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σε σχέση με τις υβριδικές απειλές και στην Ιταλία το αντιμετωπίσαμε αυτό. Η μεγαλύτερη επιχείρηση που βοηθά τις αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις πληροφοριών είχαμε μία σοβαρή απειλή σε επίπεδο κυβέρνοχώρου και σε σχέση με τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφορικής, ε, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα για την ε, προάσπιση των ε, ζήτηματων άμυνας. Τώρα σε σχέση με τη Σομαλία και το Μαλί προβάλλουμε ανθρωπιστικές ενέργειες ή και άλλες, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε και πολλούς παράνομους μετανάστες που προέρχονται από το Μαλί, την Αιθιοπία, γενικότερα από την Αφρική. Ξέρω ότι πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι για να ε, μειώσουμε αυτή τη διόγκωση της παράνομης μετανάστευσης. Αυτά σε σχέση με μία ΚΕΠΑ που θα πρέπει να είναι μία πραγματική κοινή δύναμη, ένας κοινό στρατός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την αμυντική μας ικανότητα. Δυστυχώς σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων μειώσαμε τις αμυντικές μας δαπάνες, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλό, αλλά αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Ο κύριος Κάρας. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, υπόθηκαν σχεδόν όλα. Νιώθουμε και αισθανόμαστε όλοι ότι ο τομέας αυτός ο, στο, όσον αφορά την άμυνα, την, την ασφάλεια, και ε, την έρευνα. Υπάρχουν όλες αυτές οι διαστάσεις και από αυτή την άποψη ο τομέας αυτός αφορά και την κοινωνία και την ανάπτυξη αλλά κυρίως και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αξιοπιστίας της και της αυτονομίας της. Και σύμφωνα με τις ε, μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι στόχοι που θέσαμε πριν από 10 χρόνια δεν έχουν επιτευχθεί. Αφενός μιλούμε για μια ενισχυμένη πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Από την άλλη πλευρά οι, οι εξοπλιστικές εξελίξεις, οι εξοπλισμοί στα κράτη-μέλη πραγματοποιούνται χωρίς να υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός συντονισμός και μάλιστα με προμηθευτές εκτός Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι μεμονωμένε κινήσεις ορισμένων κρατών μελών μειώνουν την ανεξαρτησία του συνόλου της Ένωσης. Άρα, μήπως θα έπρεπε να γίνει και μια συζήτηση για την μεταρρύθμιση του ε, αμυντικού κλάδου και εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκό συντονισμός στις μεταρρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζεται ότι κάθε αλλαγή θα πραγματοποιείται και θα συμβανίζει με καλύτερο συντονισμό και ποιες είναι οι προοπτικές που θεωρείτε εσείς ότι υπάρχουν, οι ευκαιρίες δηλαδή, για την οικοδόμηση μιας πλατφόρμας συντονισμού και μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας, άμυνας και έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay, Ωραία. Δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Οπότε θα συζητήσω και εγώ τον, θα πάρω και εγώ τον λόγο. Κύριε Πρέσβη, μιλούμε εδώ και αρκετό καιρό για την ανάγκη συντονισμού, για τις απαραίτητες αλλαγές και την ε, απαραίτητη αύξηση της ε, ποιότητας της παραγωγής στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Και παρόλα αυτά φαίνεται ότι τα μέσα που χρησιμοποιούμε και εμείς και τα κράτη-μέλη δεν επαρκούν, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι τα κονδύλια που δαπανούν ε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα θα πρέπει να αυξηθούν. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποιες πιστεύετε εσείς ότι είναι οι ε, προοπτικές όσον αφορά την έρευνα και την ε, εξέλιξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα ασφάλειας και Άμυνα. Και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει πολλές φορές το ε, αίτημα να ενισχυθεί η έρευνα, να ενισχυθεί η καινοτομία και ε, αναφέρομαι και στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιάννη Στόλτεμπεργκ, στο Συμβούλιο συζητήσατε μαζί του, οπότε θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να μας περιγράψετε λίγο τι συζητήθηκε. Τι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, η ανάγκη ανάληψης δράσης, οι αποστολές και στο πλαίσιο το δημοσιονομικό για το επόμενο έτος. Έχετε ε, ε απαντήσεις να μας πείτε γι' αυτό ο, ο πρέσβης. Θα μιλήσω στα γερμανικά, μιας και μου μιλήσατε γερμανικά, για την νέα ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι άλλαξε το πλαίσιο και αυτό, έχει, ε, αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή. Υπήρξαν πράγματι ε, διάφορες προσπάθειες να χαραχτεί μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι εξελίξεις από τον Δεκέμβριο του 2013, δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ΝΤΑΕΣ, το Ισλαμικό κράτος, συνέβαλαν στο ότι άλλαξε και η αντίληψη περί ασφάλισης των, των Ευρωπαίων. Σκοπός της Φεντερίκα Μεντερίνη είναι να χαραχτεί μια ευρύτατη πολιτική ασφάλειας, δηλαδή όχι μια νέα έκδοση της στρατηγικής της πολιτικής του 2003, αλλά η δημιουργία ενός νέου στρατηγικού πλαισίου, που μεταξύ άλλων θα ενισχύει και την μεταξέλιξη, ε, την περαιτέρω εξέλιξη των ε, διαφόρων ε, μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το είπε και στα κρατημέλη, το είπε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ομιλία της, ότι πρόκειται για μια συζήτηση που θα έχει ευρύ χαρακτήρα για τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, υπάρχουν, που έχουμε στη διάθεσή μας. Εδώ μιλούμε κατά κύριο λόγο για έρευνα και ανάπτυξη. Πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή. Αυτό είναι ένα ερώτημα με το οποίο ασχολείται και αυτή η Επιτροπή Προσωπικοποίητων, στην οποία συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε, η Επιτροπή αυτή δρά συμβουλευτικά προς την Κομισιόν ε, ως προς ζητήματα προϋπολογισμού και διακυβέρνησης αυτού του νέου ερευνητικού προγράμματος. Γι' αυτό άλλωστε αποκαλείται προπαρασκευαστικό μέτρο, διότι αν έχει ελεγχθεί θα μπορεί στη συνέχεια, όταν ελεγχθεί μάλλον, θα μπορέσει να μπει σε κανονική ε, γραμμή του προϋπολογισμού και αυτό θα μπορέσει να γίνει στην αναθεώρηση του ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Για το άλλο θέμα που αναφέρατε θα πρέπει να το, να το, να το δούμε. Για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα πάντως θα πρέπει να διατυπώνεται με ένα τέτοιο τρι, τρόπο ώστε όλες, όλοι οι κλάδοι και όλες οι επιχειρήσεις να μπορούν να, επο, να υποφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό. Ο κύριος Κάρας ε, ζήτησε περισσότερη συνεργασία, ρώτησε για το τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Είναι σημαντικό το ερώτημα. Τελικά η αμυντική πολιτική όμως είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Η δική μας ε, αρμοδιότητα, το δικό μας καθήκον είναι να συνοδεύσουμε, να υποβοηθήσουμε και να διευκολύνουμε την ε, συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αλλά τα κράτη-μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να δέχονται ως συντανιστή τη δική μας υπηρεσία, ούτε το ζητήσαμε ποτέ αυτό εμείς ως υπηρεσία. Το Νοέμβριο του 2014, ωστόσο, η Υπουργοί Άμυνας αποφάσισαν τη δημιουργία μιας, ε, ενός πλαισίου για τη συνεργασία στον ε, τομέα της πολιτικής άμυνας. Δεν είναι δεσμευτικό το πλαίσιο αυτό, είναι προαιρετικός ο χαρακτήρας της συνεργασίας, αλλά θα μπορούσαμε για παράδειγμα στο πλαίσιο αυτό να ζητήσουμε από την υπηρεσία να παρακολουθεί τις εθνικές στρατηγικές. Αν κάποιο κράτος μέλος, για παράδειγμα, αποφασίσει να συντάξει μια λευκή βίβλο για τη συνεργασία, η δική μας υπηρεσία θα μπορούσε να βοηθήσει. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας, παραμένει περιορισμός, περιορισμένος και η συζήτηση είναι πάντοτε πολύ ζωηρή όταν ε, αρχίζουμε να συζητούμε αυτό το θέμα και θα έχουμε την ευκαιρία το φθινόπωρο που μας έρχεται να ξανασυζητήσουμε για αυτό το θέμα. Τώρα, να απαντήσω και στα πολωνικά, γιατί ε, τέθηκαν ερωτήματα και στα πολωνικά. Πρώτα απ' όλα, για τις ε, δραστηριότητες και τα μέτρα που λαμβάνουμε κατά του δουλεμπορίου. Σωστά αναφέρατε τα νομικά ζητήματα και τα ζητήματα της έντολης. Ε, η αποστολή Uniformed, η επιχείρηση Uniformed έχει ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν δραστηριότητες ε, που έχουν αναλυφθεί στην Μεσόγειο. Ήδη πλέον τέσσερα πλοία στη Μεσόγειο, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεσή μας από κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην φάση R1 της εντολής συγκεκριμένα, που σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε μέτρα παρακολούθησης της κατάστασης. Όσον αφορά τις επόμενες ε, φάσεις, δηλαδή της σύλληψης, να το πω έτσι, των δουλεμπορικών πλοίων, για κάτι τέτοιο ε, απαιτείται απόφαση των κρατών μελών και το είπαν και ξεκάθαρα τα ίδια τα κράτη-μέλη. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια συζήτηση για το αν χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να ξεκινήσει νέα φάση ή όχι. Οι διπλωματικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη ωστόσο. Η ύπατη εκπρόσωπος έχει κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και αποστολές και στην Αφρική και έχει δηλώσει ότι δεν, δεν εξαντλείται εκεί η στρατηγική μας στην Αφρική. Είναι ένα, τμήμα της και μόνο. Επίσης υπάρχουν δραστηριότητες στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έγιναν συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα Μίλησε επίσης μαζί η ύπατη εκπρόσωπης με τον, ε, με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ και στο Λουξεμβούργο. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας <clears throat> δεν μπορώ να πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ε, πολύ έντονες εργασίες, αλλά αυτό ε, σχετίζεται και με τις επιμέρους πτέρυγες και μερίδες κρατών στο Συμβούλου Ασφαλείας και στον ΟΗΕ ευρύτερα. Πάντως μπορούμε να μιλήσουμε για, έναν για μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Με άλλα λόγια αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς ε, αναπτύσσουμε τις ε, δραστηριότητες μας, τις διπλωματικές, Υπάρχει και ένας Ιταλός αξιωματούχος ο οποίος συναντάται σήμερα στη Νέα Υόρκη με τη γραμματεία του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα μας ενημερώσει, θα μας απαντήσει και σε διάφορα ερωτήματα και όλα αυτά θα γίνουν στις 31 Ιουλίου, δηλαδή πριν τη διακοπή για το καλοκαίρι. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά κονδύλια ε, για την άμυνα, αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις από το έτος 2007 ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, δηλαδή έτσι όπως ε, αναφέρονται συγκεκριμένα ως κοινέ δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ε, επιτύχει κάποιες, κάποια εξαιρετικά αποτελέσματα. Ακόμη ούτε μπορεί έτσι απλά να μετουσιωθούν ε, σε διεθνείς υποχρεώσεις γιατί ακριβώς είναι αρμοδιότητα των ίδιων των κρατών μελών και γι' αυτό ε, μιλούμε πιο πολύ για προπαρασκευαστικά μέτρα και για ερευνητικά προγράμματα. Το ερευνητικό πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο να χρηματοδοτηθεί ε, με υψηλότατα ποσά αλλά ε, είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον που έχουμε καθιερώσει συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Είχαμε τη δυνατότητα και από το πρόγραμμα πλαίσιο και από τον, από τον ορίζοντα 2020 να λάβουμε κάποια μέσα χρηματοδοτικά ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, τη διπλή χρήση, τα προϊόντα διπλής χράσης, αλλά ε, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, μας έχουν, έχουν συμβάλει στην δημιουργία ε, αυτού του ερευνητικού προγράμματος. Τώρα, για τον Γενικό Γραμματέα δεν συμμετείχα που, και το Συμβούλιο εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν συμμετείχα στη συζήτηση. Επικεντρώθηκαν λόγω του περιορισμένου χρόνου σε ε, τα σημαντικότερα ζητήματα ήταν κάπως επιτελική η συζήτηση δηλαδή επικεντρώθηκε στις ε, επιχειρήσεις άλλωστε η κυρία Μογκερίνη ήταν και εκείνη προσκεκλημένη των Υπουργών Άμυνας ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η δυνατότητα επέμβασης, παρέμβασης και πώς θα ενισχυθούν αυτές ε, τώρα για το τι κάνει το ΝΑΤΟ Υπάρχει βεβαίως αυτός ο χαρακτήρας και η ευρωπαϊκή διάσταση ακόμη και όταν ε, δραστηριοποιούμαστε στο Αφγανιστάν στη Μέση Ανατολή και αυτό είναι και προς όφελος του ίδιου του ΝΑΤΟ διότι από την σύνοδο ε, κορυφή στο Βάλι το ΝΑΤΟ εμείς μάλλον επικεντρωνόμαστε στις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 Υπάρχει δηλαδή, μπορώ να σας πω πάντως, μια ε, πολύ φυσική και αγαστή συνεργασία και συμπληρωματικά ε, μέτρα λαμβάνονται. Τις άλλες ερωτήσεις θα τις απαντήσω στα αγγλικά. Η οικονομική διάσταση της ε, βιομηχανίας άμυνας. Έχετε δίκιο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός τομέας της ευρωμαϊκής Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Άμυνας γενικά. Μιλάμε για 800.000 θέσεις εργασίας. Δεν μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά φυσικά υπάρχει μια βιομηχανία μεγάλη, μικρή. Ξέρουμε ποιες είναι οι μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν και πολλές ΜΜΕ που απασχολούνται στον τομέα αυτό. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία τους. Συμφωνώ βεβαίως ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ποιότητα. Και όταν δείτε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιαίτερα από αυτά που καθοδηγούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ή τη δημιουργία δορυφόρων, επικοινωνίας μέσω δορυφόρων, αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε σε μια ευρωπαϊκή αυτονόμηση για να αναπτύξουμε ικανότητες και να μην τις ε, προμηθευόμαστε από άλλους. Όπως ισχύει με τα μη επανδρομένα οχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε νέα προγράμματα όποτε τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα για κάτι τέτοιο, γιατί ε, ξέρετε ότι η πολιτική άμυνας είναι εθνική. Άρα αν μιλάμε για ασφάλεια και άμυνα στον ε, κυβερνοχώρο ή στις ε, θαλάσσιες μεταφορές, θα πρέπει να το δούμε με τα κράτη-μέλη. Μίλησα για το στόχο 2% του ΑΕΠ. Αυτός είναι ένας στόχος του ΝΑΤΟ. Δεν θέλω να τον σχολιάσω γιατί δεν είναι δική μας ε, δέσμευση. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να επιταχύνουν και να φτάσουν στο στόχο το νωρίτερα. Αν μπορούν να το κάνουν μας ε, πληροφορούν επ' αυτό, αλλά δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην ε, Πολωνία, στις Βαλτικές χώρες και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει προωθηθεί αυτή η θέση. Και αν το δούμε από πλευράς ευρωπαϊκής προοπτικής είναι κάτι το θετικό. Τώρα, ως προς τον συντονισμό μεταξύ εθνικών ενόπλων δυνάμεων και της, ε, των εθνικών πολιτικών άμυνας ε, δεν μπορούμε παρά να το ενθαρρύνουμε γιατί μιλώ για εθελούσια βάση συνεργασίας σας το προανέφερα αυτό για πολλούς λόγους, αλλά ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσον. Δεν θέλουμε να το επιβάλλουμε σε κάποια χώρα να συνεργάζεται με τους πάντες, αλλά αν υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα σε περιφερειακό επίπεδο, αυτό μπορεί να το προωθήσει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Ένα παράδειγμα είναι στο Eindhoven ε, που πρόθεσε ένα νέο σχέδιο, δηλαδή έξι κράτη-μέλη έχουν ε, δημιουργήσει μία συνιστόσα ως προς την, στις εναέριες μεταφορές και τους αεροδιαδρόμους. Όποιος θέλει λοιπόν να μεταβεί στο Μάλι για ανθρωπιστική βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο, έρχεται σε επαφή με το Eindhoven, το οποίο και προωθεί αυτούς τους αεροδιαδρόμους. Εγώ επισκέφτηκα αυτό το κέντρο. Είναι μία συνεργασία που θα πρέπει να προωθήσουμε. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια είναι τα ευεργετήματα. Σε σχέση τώρα με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η εντολή μας είναι περιορισμένη γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αλλά μιλάμε για προστασία των ήδη υπαρχούσων αποστολών, γιατί δεν έχουμε ένα ευρωπαϊκό project για την ασφάλεια στον κυβέρνοχώρο. Το ΝΑΤΟ έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά είναι μία συμμαχία άμυνας, άρα είναι διαφορετικό. Τώρα όμως που θα προωθήσουμε αυτή την ε, πολιτική πλαίσιο, για να αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές θέλουμε να δούμε και το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τώρα, ως προς τις αποστολές μας στο Μαλί και τη Σομαλία, υπάρχουν πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές ως προς τις στρατιωτικές αποστολές τι κάνουν στην ουσία εκπαιδεύουν το στρατό στο Μαλί και στη Σομαλία Πρόκειται για αποστολές εκπαίδευσης και παροχή σύμβουλων. Όμως στο Σαχέλ έχουμε μια πολιτική φύση συνεργασίας στο Μαλί και στο Νίγηρα, καθώς και στο Σαχέλ. Και είπαμε στα κράτη ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ικανότητά τους για να καταπολεμήσουν την ε, παράνομη μετανάστευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι διώκουμε τους μετανάστες, πρέπει να τους προστατεύσουμε. Όμως μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με αυτές τις υπηρεσίες στο Νίγηρα και στο Μάλι για να είναι πιο αποτελεσματικές. Ένα λοιπόν από τα μέτρα που δεν έχει καταγραφεί και τόσο πολύ γιατί ε, μιλήσαμε για την θαλάσσια αεροπειρατεία είναι η συνεργασία σε μια πόλη στον Νίγηρα στα σύνορα με τη Λιβύη. Εκεί εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε επιτοπίως με τις αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις χωροφυλακής του Νίγηρα για να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές ροές, διότι ο Νίγηρας και όλη η περιοχή του Σαχέλ είναι ε, ένα ε, σημείο, ένα κόμβος, ένα κομβικό σημείο διέλευσης. Γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε εκεί για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις ε, ροές αυτές. Και από τότε που προωθήσαμε αυτή την αποστολή, αν και είμαστε στην πρώτη φάση της ε, θαλάσσιας αυτής ε, αποστολής, τα τελευταία στοιχεία είναι ενθαρρυντικά γιατί βλέπουμε ότι λιγότεροι μετανάστες επιβιβάζονται στα πλοία και δεν έχουμε και τόσους θανάτους, ευτυχώς. Βεβαίω οι διακινητές γνωρίζουν ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι που προωθούν αυτή την ε, θαλάσσια αποστολή και κάπως αποθαρρύνονται. Όπως ε, και η Frontex που είναι μια πολιτικής ε, φύσης συνεργασία και όχι στρατιωτικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρέσβη. Έχουμε λίγο χρόνο αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις επί του θέματος. Άρα μπορούμε να έχουμε και ένα δεύτερο γύρο, αν, αν το επιθυμούν τα μέλη. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον πρεσβευτή μετά το θέμα μετά την ε, νέα θαλάσσια αποστολή στη Μεσόγειο. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι τρόποι για να ερμηνεύσουμε την εντολή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών ή των ψηφισμάτων γενικότερα. Μιλάμε για μια πρώτη φάση της εντολής και συμφωνώ ότι η παρουσία μας ε, κάθε αυτή αφορά το, την εποπτεία της ε, δραστηριότητας στη Μεσόγειο. Τη μετανάστευση, τις ε, μεταναστευτικές ροές μέσω Μεσογείου. Έχουμε ένα μέσο αναχέτησης ή πρέπει να το συνδέσουμε με άλλες προσπάθειες, άλλες επιτόπιες ε, προσπάθειες στην ε, Βόρειο Αφρική. Και ίσως θα πρέπει να είμαστε και πολύ σύντομοι, να αποτιμήσουμε δηλαδή την επόμενη φάση. Εντάσσεται στο... στην παρούσα εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ποιο θα είναι το επόμενο ψήφισμα. Και ενισχύοντας το θέμα της δημοσιονομικής πτυχής, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες προκλήσεις ανά τον κόσμο μετά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και νομικής ε, υφής ε, ζητήματα για να δούμε πώς ε, θα μπορέσουμε να δράσουμε περαιτέρω. Ο περιορισμός της θαλάσσιας επιχείρησης ίσως μας επιβληθεί και από τα δημοσιονομικά μας. Ποια είναι η εξισορρόπηση μεταξύ στόχων αναγκαιότητας, αποδοτικότητας και οικονομικών. Έχετε δίκαιο, υπάρχουν περιορισμοί δημοσιονομικής υφής το θέμα της χρηματοδότησης των αποστολών είναι ένας ε, τομέας όπου δεν έχει επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος από το 2013 και μετά. Προσπαθήσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με βάση αυτό τον μηχανισμό ε, Αθηνά, Αθήνα Mechanism, και συνεπώς αυτή η θαλάσσια επιχείρηση χρηματοδοτείται από τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη με κοινό κόστος, το οποίο δεν είναι υπέρογκο. Βασιζόμαστε από τα κράτη-μέλη τη χρηματοδότησή τους. Ε, ως προς την αποστολή, υπάρχει αυτό το θέμα της νομικής ασάφειας, η διατύπωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα και αν έχουμε εντολή. Δηλαδή πολλές φορές μιλάμε για καταστροφή πλοίων, αυτό δεν έγινε δεκτό. Μιλάμε για κατάσχεση και διάθεση ε, πλοίων, αλλά θα πρέπει να το συμφωνήσουμε. Η διοίκηση ε, έλαβε υπόψη τα λιμάνια αποβίβασης, αλλά χρειαζόμαστε φυσικά και άδεια για την κατάσχεση των πλοίων και τη διάθεσή τους. Εάν μιλάμε για τους διακινητές, οπωσδήποτε θα πρέπει να δικαστούν κάπου, είτε στη χώρα προέλευσης, είτε στη χώρα που θα τους δεχτεί. Άρα υπάρχει κάποια ομοιότητα με τη δράση μας στο κέρας της Αφρικής. Δηλαδή, όταν συλλαμβάνουμε τους πειρατές πρέπει κάτι να τους κάνουμε. Άρα έχουμε συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες που τους δέχονται και τους δικάζουν, όπως ε, ίσχυσε με την περίπτωση του Μαυρικίου. Ως προς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, βεβαίως είμαστε φιλόδοξοι, οι περισσότερες επιχειρήσεις μας είναι πολιτικές, όπως αναφερθήκατε στο κοσυφοπέδιο, και η γραμμή του προϋπολογισμού ε, της ΚΕΠΑ έχει μία οροφή. Άρα δεν θα επαυξηθεί φέτος, καλά κρατούμε, αλλά αν πρέπει να κάνουμε κάτι το καινούριο, κάτι της εμβέλειας, ας πούμε, της ανάλογης επιχείρησης στο κοσυφοπέδιο. Δεν υπάρχουν σχέδια, αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας. Αυτό θα είχε επίπτωση στον προϋπολογισμό φυσικά. Το συζητήσαμε με την Επιτροπή και είπα ότι εκπρόσωπος το ΙΔ ε, με τους επιτρόπους που ασχολούνται με θέματα εξωτερικής πολιτικής για να μην ε, φτάσουμε δηλαδή ακόμα και κάτω από το κατόφλι μας ως προς τις δυνατότητες ε, δαπάνης, διότι αυτό θα μας ε, περιόριζε ως προς τις ε, πολιτικές μας δραστηριότητες ε, της ΚΕΠΑ. Και κάτι άλλο που ανέφερα πριν, το ενδιάμεσο, την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολετού σχεδίου. Και αυτό θα μας απασχολήσει μελλοντικά. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Να σας ευχαριστήσω και για την παρουσίαση. Παρακαλώ. Κύριε Κόλλον, κύριε Βαλάρη. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Πρώτον, να μας πείτε για τα μη επανδρομένα σκάφη. Ξέρουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους ε, μηχανήματα. Και οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, για τους αερολιμένες. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι λοιπόν. Και βεβαίως πέρα από την στρατιωτική χρήση αυτών των μηχανημάτων που εξετάζεται και σε διεθνές επίπεδο. Πού βρισκόμαστε λοιπόν. Και δεύτερον, είπατε ότι προσπαθούμε να διαχειριστούμε ε, όλο αυτό το, κύμα μετανάστευσης. Τι κάνουμε στο άλλο άκρο. Τι συμβαίνει, τι κάνουμε για την, ε, για την αντιμετώπιση των ε, αιτίων, των ανισοτήτων και των αδικιών για να μην έρχονται οι άνθρωποι αυτοί. Κύριε Βαλέρα, θα μιλήσω και πάλι σου ειδικά. Βάλετε παρακαλώ τα ακουστικά σας, γιατί δεν θα με καταλάβετε αλλιώς. Είπατε λοιπόν ότι δεν γίνεται πολύς λόγος για την μείωση της, ζήτησης. Εγώ νομίζω ότι ακριβώ αυτό ήταν το θέμα της συζήτηση μεταξύ των Υπουργών και μάλιστα ότι ζητήθηκε να ότι πρέπει να αναλυθούν δράσεις για, την, για τη βήθηση πλοίων. Μιλήσαμε και για τα PNR, ε, για την ανάγκη να δοθεί γρήγορα μια απάντηση ε, στα προβλήματα χωρίς ωστόσο να εξεταστεί αν όλα αυτά συμφωνούν με, τις, με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Πολλές φορές δηλαδή έχουμε την αίσθηση ότι το Συμβούλιο των Υπουργών επιδεικνύει μια βιασύνη να ε, επιδείξει και να καταλήξει σε θέση και να επιδείξει στους πολίτες ότι αναλαμβάνονται και δράσεις για να προστατευτούν οι πολίτες αλλά πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και για μένα ως ευρωβουλευτή αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Το να εργάζομαι δηλαδή και να εργαζόμαστε σε τέτοιες συνθήκες όπου το Συμβούλιο των Υπουργών εκδίδει διακηρύξεις και δηλώσεις οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι καν εκτελέσιμες. Ε, κύριε Πρέσβη, για τα μη επανδρομένα σκάφη δεν έχουμε συγκεκριμένη πολιτική για τα μηχανήματα αυτά. Ίσως ενδεχομένως επειδή είναι καινοφανές ε, φαινόμενο. Ε, σίγουρα όχι στο στρατιωτικό τομέα πάντως. Η δουλειά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικεντρώνεται στην τεχνολογία την ανάπτυξη δηλαδή μιας ευρωπαϊκής τεχνολογίας για την κατασκευή μη επανδρομένων ε, ε, αεροσκαφών, ώστε να μπορούμε να κατασκευάσουμε τέτοιου είδους μηχανήματα αν χρειαστεί. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πώς θα ε, εξασφαλίσουμε ότι η χρήση των σκαφών αυτών θα είναι ασφαλής στον εναέριο χώρο. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και για τη διαχείριση του συστήματος Caesar. Πάντως βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτή η δουλειά. Πάντως έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις του διεθνούς δικαίου ή από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου για την μεταναστευτική κρίση. Φυσικά, τα αίτια είναι σημαντικότατο ζήτημα και είπατε εκπρόσωπος ε, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι μία μόνο διάσταση και δεν είναι η απάντησή μας. Γιατί έχουμε χώρες προέλευσης, χώρες ε, ε διέλευσης και γι' αυτόν τον λόγο ε, το Νοέμβριο θα διοργανωθεί και στη Μάλτα μια σύνοδος κορυφής με αφρικανικές χώρες και θα ε, θα προσπαθήσουμε να ανακατευθύνουμε και ορισμένα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και βοήθεια προς την ε, οικοδόμηση θεσμών στην Ιγυρία και σε άλλες χώρες, προκειμένου να μπορέσουν αυτές οι χώρες να αναπτύξουν δικαστικά συστήματα και να ανακοπεί και με αυτόν τον τρόπο ε, το μεταναστευτικό κύμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο δική μας αρμοδιότητα, ούτε εμείς μόνο μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα με πλοία, όταν, το, όταν οι μετανάστες έχουν ήδη φτάσει στη θάλασσα. Και για την ερώτηση της κυρίας Βαλέρο. Ε, είναι αλήθεια ότι η εικόνα ε, είναι σημαντική. Εμείς όμως ε, λέμε το εξής, ότι η απόφαση για την ε, πραγματοποίηση της ε, επιχείρησης δημιουργήθηκε πολύ προσεκτικά, συντάχθηκε πολύ προσεκτικά και αυτό που εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης. Επίσης έχουμε αναλάβει και κάποιες ε, διπλωματικές ενέργειες στη Γενέβη, για παράδειγμα. Ε, μιλήσαμε με τον ύπατο εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και του εξηγήσαμε ε, τους, ε, τις δικές μας νομικές ε, υποχρεώσεις σύμφωνα με, τους, με το διεθνές δίκαιο ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλα των, όλων των μεταναστών. Όταν για παράδειγμα φτάνουν στην στεριά ε, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάζουμε τα αιτήματα ε, ασύλου τους. Γιατί, ε, και είναι περίπλοκο αυτό το ζήτημα, γιατί πρέπει σε εκείνη την φάση να εξετάσει κανείς ποιος είναι οικονομικός μετανάστης, ποιος είναι πρόσφυγας. Πάντως συνεργαζόμαστε και με άλλες υπηρεσίες, με τη Europol, με τη Frontex. Θα και σας διαβεβαιώ ότι εμείς θα ενισχύσουμε τις δικές μας αποστελές ε, στην ε, Βόρεια Αφρική, στην Υποσαχάρια Αφρική προκειμένου να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ποπόφσκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζουμε να παρευρεθείτε και πάλι σε μια επόμενη συνεδρίασή μας ε, και Τώρα που έχει ολοκληρωθεί και αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ένα μικρό διάλειμμα να κάνουμε. Παρακαλώ να επανέλθουμε 10.30 ακριβώς, γιατί θα αρχίσουμε τη δημόσια ακρόασή μας για τον έλεγχο για τις εξαγωγές όπλων. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Παρακαλώ να είστε πίσω εγκαίρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ladies uh, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Καθίστε. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση μας. Ε, πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας, που είναι η δημόσια ακρόαση για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ε, ομιλητές μας. Ο πρώτος είναι ο Πιέγα Γνώλοτο ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, ε, Δράσης ε, και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τον έλεγχο των εξαγωγών των όπλων στο Συμβούλιο. Θα μας πει ορισμένα πράγματα για τη, τη, τη σχέση της ομάδας αυτής εργασίας και της δουλειάς της στο πλαίσιο της ΕΕΔ. Ο δεύτερος ομιλητής μας ε, εκπροσωπεί το Safe World, ε, μία μη κυβερνητική οργάνωση και ο, τρί, ε, ο τρίτος ομιλητής μας, ο κύριος Γιάν Πίε, από την ε, αεροναυπηγική και από τον, την Ένωση ε, Αεροναυπηγικής και Διαστημικών Υπηρεσιών ε, που είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης στο πλαίσιο του ελέγχου των όπλων Δεσμευτικό είναι το κείμενο της κοινή θέσης για ε, τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποβάλει αιτήσια ε, έκθεση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η εισηγήτριά μας είναι η κυρία Μπότλ Βαρέρο ε, και η δημόσια αυτή ακρόαση γίνεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προετοιμασίας για αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, πρώτα ο κύριος ε, Λωτών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την ευκαιρία να ε, σας παρουσιάσω τις εργασίες της ΚΟΑΡΜ και να σας πω σε ποιο επίπεδο θεσμικό εξελίσσεται. Το COARM είναι ε, η ομάδα ε, εργασίας, μία από τις πολλές του Συμβουλίου, ε, που ασχολείται με το θέμα των συμβατικών όπλων. Ξέρετε ότι υπάρχει και η Κορεπέρ και υπάρχει και στο υψηλότερο επίπεδο το Συμβούλιο Υπουργών. Η COARM είναι υπεύθυνη για τις εξαγωγές των συμβατικών όπλων υλικών συστημάτων ε, και οι ομάδες εργασίας που έχουν να κάνουν ε, με την ΚΕΠΑ, μεταξύ, μεταξύ των οποίων και η ΚΟΑΡΜ που έχει να κάνει με την Αφρικανική Ένωση, μια άλλη με την Ασία, είπα, ε, ο επικεφαλής είναι ο εκπρόσωπός μας στην ΑΕΔ είμαι εδώ ως ε, εκπρόσωπος μίας από τα, ε, ενός από τα τμήματα ε, που εκπροσωπούνται στην ΕΙΕΔ. Υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο, όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, ε, που είναι η κοινή θέση 2008 944 που εγκρίθηκε ε, το 2008 και όπως γνωρίζετε αυτή η κοινή θέση ουσιαστικά έρχεται μετά από τον ε, κώδικα δεοντολογίας για τα όπλα. Από τον κώδικα δεοντολογίας μέχρι την κοινή θέση ο στόχος παραμένει ίδιος, είναι η προώθηση σύγκληση των κρατών ε, μελών και των πολιτικών τους ε, για τις εξαγωγές των όπλων. Σύγκληση, η ε, υποστήριξη της σύγκλησης, αυτό είναι το κλειδί των εθνικών πολιτικών εξαγωγών όπλων με ένα υπόβαθρο που δεν έχει αλλάξει και που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το πλαίσιο. Ξέρετε ότι είναι μια εθνική αρμοδιότητα, τα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει ότι υπάρχει μια σύγκληση, ένα πλαίσιο σύγκλησης και ένας μηχανισμός σύγκλησης, όμως σε τελική ανάλυση παραμένει μια εθνική ευθύνη το θέμα αυτό. Τώρα, ε, πώς ε, υποστηρίζεται αυτή η σύγκληση ε, σε, τέσσερα, σε τέσσερις πτυχές βασίζεται, είναι τα κοινά κριτήρια. Υπάρχουν οχτώ κριτήρια στην κοινή θέση που είναι τα ελάχιστα ε, βάσει των οποίων το τα κράτη-μέλη πρέπει να αξιολογούν ε, τις εθνικές πολιτικές εξαγωγών τους που καλύπτουν μια ευρία κλίμακα εξωτερικής πολιτικής, θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Αυτό είναι η Πρώτη πτυχή. Δεύτερη πτυχή, ε, όταν μιλάμε για τα όπλα, μπορεί να σας φαίνονται απλά τα πράγματα, αλλά το πεδίο ε, εφαρμογής των συνθήκων για τα ε, όπλα είναι πολύ ευρύτερο. Υπάρχουν ε, πολλές, πο, εξοπλισμός που έχει να κάνει με τις επικοινωνίες, με την επιμελητεία και αναφέρεται σε, μια, σε έναν κατάλογο κοινό στρατιωτικό που συμπεριλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο για το θέμα αυτό. Τρίτη πτυχή είναι ανταλλαγή απόψεων ε, για ε, πληροφορίες ε, και ανταλλαγή απόψεων. Η ΚΟΑΡΜ συνεδριάζει μία φορά το μήνα και τα κράτη-μέλη εκεί μπορούν να συζητήσουν την αξιολόγηση της ασφάλειας σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προ... προορισμό, πάντοτε χάριν σύγκλησης, όπως είπα και προηγουμένως. Και τέλος, τελευταία διάσταση είναι ε, ένας ε, μηχανισμός ε, αξιολόγησης και διαβούλευσης. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διαβουλεύονται και να συμβουλεύονται το ένα το άλλο όταν πρέπει να γίνει μία αδειοδότηση για μία συναλλαγή την οποία έχει απορρίψει ένα άλλο κράτος μέλος προηγουμένως με σκοπό και πάλι την ανταλλαγή απόψεων. Αν υπάρχει ένας καλός λόγος για να αρνηθεί ένα κράτος μέλος μία συναλλαγή πρέπει να το γνωρίζουν αυτό τα υπόλοιπα κράτη-μέλη όταν πρόκειται να γίνει μια παρόμοια συναλλαγή, ώστε να μπορεί το κράτος μέλος ε, εν προκειμένου να, να καταλήξει στην ίδια αρνητική αξιολόγηση της συναλλαγής αυτής. Και για να ολοκληρώσω ε, το, το, το παζλ της ε, ε, κοινής θέσης περιλαμβάνει μία βασική απέτηση ότι κάθε χρόνο πρέπει να παρέχουν δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη προκειμένου να προετοιμάζουν και να δημοσιεύουν ε, την ετήσια έκθεση για τις εξαγωγές όπλων. Αυτό είναι ε, ο βασικός μηχανικός ε, βάσει του οποίου και η ε, κοινωνία των πολιτών αλλά και τα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να γνωρίζουν τι γίνεται σε σχέση με μια συγκεκριμένα συγκεκριμένο προορισμό βάσει των αριθμητικών στοιχείων που βλέπετε στον κατάλογο κάθε φορά και βάσει επιπλέον πληροφοριών όπως ε, οι διαβουλεύσεις ε, στις οποίες προβαίνουν τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένους προορισμούς. Όσον αφορά τώρα την αναθεώρηση της κοινή ε, θέσης, ήταν επίσης ε, ένα προαπαιτούμενο το 2008 ότι κάθε τρία χρόνια ε, μετά την έγκρισή της πρέπει να αναθεωρείται και αυτό έχει γίνει το 2012 και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της αναθεώρησης αναφέρθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της, ή, του Νοεμβρίου του 2012 και εξολόγηση των κρατών μελών του Συμβουλίου τότε ήταν ότι ε, ακόμη ότι ήταν θετική αξιολόγηση ότι μπορεί να υποστηρίξει τη σύγκληση, όμως πρέπει να γίνει περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή την εφαρμογή των τεσσάρων ε, ε, πτυχών που προσπάθησα να συνοψίσω προηγουμένως, ε, ειδικότερα την άρνηση, την έγκαιρη προειδοποίηση που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, να είναι πιο φιλικά προς το χρήστη, να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες κλπ και τα τελικά συμπεράσματα του Συμβουλίου που έχουν ε, να κάνουν ε, με αυτές τις βελτιώσεις ε, της εφαρμογής από το 2012 και εξής. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο έλαβε υπόψη η αναθεώρηση είναι ένα τη της συνθήκης για το εμπόριο όπλων. 26 από τα 28 μέλη της Ένωσης την έχουν επικυρώσει, όλα τι έχουν την υπογράψει. Ε, και αυτό που κάναμε εμείς στο ΚΟΑΡΜ, ε, αλλάξαμε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές μας για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε κάποιους υπεύθυνους εθνικής αδειοδότησης ώστε να μπορούν οι γενικές αυτές κατευθυντήριες γραμμές να συνάδουν και με την κοινή θέση αλλά και με τις εθνικές στρατηγικές. Ε, να σας ε, ενημερώσω επίσης ότι δεν έχουμε ε, μία ε, νέα θέση. Εξακολουθεί να υφίσταται η κοινή θέση του 2008. Ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε βελτιωμένες ε, κατευθυντήριες γραμμές στο μέλλον, ε, πιο αποτελεσματικές, καλύτερα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ελπίζουμε και μία νέα πλατφόρμα η οποία θα μας δώσει περισσότερες δυνατότητες. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει και εκείνο να γνωμοδοτήσει για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκληση στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λωτό. Ε, Ο κύριος Ίσμπης από τη Safer World, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παραβρεθώ εδώ όπως αναφέρθηκε. Εργάζομαι για την οργάνωση Safer Wall, που είναι ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός ε, για την ε, αποτροπή συγκρούσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας της ζωής. Εγώ είμαι επικεφαλής του τμήματος ε, φορητών όπλων και συμβατικών όπλων και το εμπόριο αυτών. Η υπόθεση που θα σας, παρουσιάσω σήμερα είναι ότι το σύστημα μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσει και χρειάζεται να βελτιωθεί, ενδεχομένω να τροποποιηθεί και ελπίζω ότι θα σας πείσω ότι έχω δίκιο στην υπόθεση μου αυτή. Για να επανέλθω λίγο σε αυτό που ε, αναφέρθηκε για το, ε, το ιστορικό και να συμπληρώσω αυτό που είπε και ο Διάνο, Αν δείτε λοιπόν το πώς βρεθήκαμε στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα, θα συμφωνήσω κι εγώ ότι η ανάπτυξη, η, κατάσταση, η κατάρτιση ενός ενωσιακού συστήματος είναι ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Αν πάμε στο παρελθόν, θα δείτε ότι υπήρχε ένας συνδυασμός ε, διαφόρων πραγματικοτήτων, υπήρχε ψυχρός ε, ψυχρός πόλεμος, ε, υπήρχε ένα μυστικό εμπόριο ε, και όλα αυτά έφεραν πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Και αυτό φάνηκε και στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Ο οποίος άλλωστε συνέβαλε κιόλας σε αυτήν την νέα φάση όταν τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και ανέλαβαν δράση και έτσι υπήρξε μια μετάβαση προς ε, γενικά, ε, γενικούς κανόνες όσον αφορά το εκτιμόμενο αποτέλεσμα ε, μιας μεταφοράς. Ήταν μια ριζική αλλαγή αυτή στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Η Safer World υποστηρίζει στεναρά το υπάρχον σύστημα. Όχι απαραίτητα σε όλες τις περιπτώσεις την εφαρμογή του, αλλά σίγουρα τη βασική ιδέα στην οποία βασίζεται το σύστημα. Ωστόσο, ε, αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι ενδεχομένως ε, απαιτείται η νέα φάση, μια νέα φάση, μια νέα μετάβαση. Και να σας υπενθυμίσω ε, ένα σχόλιο που έκανε ένας ένας αξιωματέχος της COARM ότι η, ελ, η έλεγχη εξαγωγές όπλων είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη δικασία. Τα κριτήρια που αναφέρθηκαν είναι βασικά τα ίδια ε, που υπήρχαν και στον κώδικα διοντολογίας του 98 μπορεί κανείς να, ε, να ε, επιστρέψει ακόμη και στα αντίστοιχα κριτήρια του Λουξεμβούργου το 1991 και της Λισαβόνας το 1992, θα δείτε ότι η φύση των ε, κριτηρίων δεν έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε, ενώ ο κόσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αλλάξει δραματικά από το 1991 και το 1992. Οπότε υπάρχει το ερώτημα αν το σύστημα έχει συμβαδίσει και με τις αντίστοιχες αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει. Αν δηλαδή και η, ε, ενώ, ε, υπήρχε το 91 τουλάχιστον ε, ένα κλίμα ε, αμοιβαίας επιφυλακτικότητας όταν έρχονταν στην GoArm τα παλιά χρόνια, το 91 ε, συνέρχονταν σε συνεδριάσεις οι αξιωματούχοι της GoArm και δεν αντάλλασαν καν απόψεις γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η επιφυλακτικότητα μεταξύ των κρατών μελών. Έχουν λοιπόν υπάρξει έκτοτε προσπάθειες για την αναθεώρηση και την ε, τροποποίηση του συστήματος, ε, αλλά φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια ε, πολύ δύσκολη φάση Λοιπόν, ο κώδικας δοντολογίας ε, συμφωνήθηκε και υπερψηφίστηκε το 1998 και υπήρξε και δεσμευτική απόφαση το 2008, ε, πολιτική απόφαση πλαίσιο, αλλά όπως είπα επί της ουσίας δεν έχουν υπάρξει ουσιώδεις αλλαγές. Και όσον αφορά την αναθεώρηση της κοινή θέσης, Εμένα με εξέπληξε το γεγονός ότι στην πράξη η αναθεώρηση διαπίστωσε ότι η διατύπωση της κοινή θέση ήταν τέλεια και δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Και στη δεύτερη φάση στην οποία αναφέρθηκε και ο πιάνο, ε, φάνηκε ότι, ότι υπήρξαν αλλαγές, ίσονος σημασίας όμως που επικεντρώθηκαν κυρίως στο να ε, ε, ευθυγραμμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη για, την, για το εμπόριο όπλων. Ε, αφορά βεβαίως και τους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων, θετικότατο βήμα αυτό, αλλά όσον αφορά τα κριτήρια, εξέτασε σε βάθος μόνο δύο κριτήρια. Και ένα από το, ε, το κριτήριο μάλλον στο οποίο επικεντρώθηκαν συζητήσεις ήταν το 7 όσον αφορά την την απόκληση. Και το ζητούμενο σε αυτό το κριτήριο είναι πώς, ποια είναι η ελληνεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών με τρίτες χώρες και όχι τόσο ε, ε, να εξεταστεί αν θα πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά των ίδιων των ευρωπαϊκών κρατών. Η κοινή θέση συνέπεσε συμπτωματικά με την Αραβική Άνοιξη. Εγώ θεωρήσα ότι αυτό θα ήταν μια αφορμή για τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε βαθιές αλλαγές. Αν και πρέπει να πω ότι έκτοτε δεν έχω δει τις αλλαγές αυτές που ανέμενα, ούτε στο σύστημα ούτε στην πράξη. Το 2010 λοιπόν υπήρχαν 8,25 ε, δισεκατομμύρια ε, άδειες ε, σε αξία. Αυτές αυξήθηκαν σε 9,5 δισεκατομμύρια, 26 10% επί του συνόλου δηλαδή. Και το 2013 το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο αδειών ανήλθε σε 10,75 δισεκατομμύρια. 29% του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου Και αυτό που βλέπουμε με την ε, σαουδική επέμβαση στην Ιεμένη είναι ότι παρά την ε, ανθρωπιστική κρίση και κάποιες αμφιλεγόμενες τακτικές που ακολουθήθηκαν, η, η, τροφοδοσία ε, στρατιωτικού εξοπλισμού προς τους ε, συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας φαίνεται να συνεχίζεται όπως και πριν. Και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ε, πρόσφατα άδεια για βόμβες και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και μια αντίστοιχη άδεια, θα εκδοθεί μια αντίστοιχη άδεια πολύ σύντομα. Τέλος πάντων, το σύστημα έχει προβλήματα. Ποια είναι η δομή του, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί. Ε, κάπως το έπιασε το θέμα αυτό και ο Πιάνο. Υπάρχουν τέσσερα κριτήρια με βάση τα οποία κανείς αξιολογεί αν, πιστε, αν αξιολογεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για παραβιάσεις, ε, απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, τότε απλά ε, δεν εκδίδει την άδεια. Υπάρχουν άλλα τέσσερα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σε αυτά ε, συγκαταλέγονται ε, ή ο κίνδυνος εκτροπής, η συμπεριφορά απέναντι στο διεθνές δίκαιο κτλ. Ε, κάθε μεταφορά αξιολογείται και κρίνεται κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι για την τρομοκρατία ή προς το διεθνές δίκαιο και έτσι εκτιμάται η χώρα συνολικά. Οι κίνδυνοι δηλαδή που συνδέονται με κάθε μεταφορά. Και βεβαίως έχουν γενική ισχύ τα κριτήρια αυτά. Όλα τα ε, κράτη παραλαβής ε, θα πρέπει να αντιστοιχούν και να πληρούν ε, τα ίδια, τις ίδιες προδιαγραφές. Ένα από τα κριτήρια, το 5 συγκεκριμένα, σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Είναι ένα κριτήριο που επιτρέπει την μεταφορά ε, ε, αν πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, τότε επιτρέπεται η έκδοση άδειας. Επίσης, μπορούν να ληφθούν υπόψη οικονομικά συμφέροντα, εμπορικά συμφέροντα, αλλά αυτά δεν θα πρέπει να υπερισχύουν ή να αντίκεινται σε κάποια από τα υπόλοιπα κριτήρια. Άρα βασιζόμαστε στον κίνδυνο. Ποιες είναι οι πιθανότητες κάτι να πάει στραβά στο μέλλον. Πού λοιπόν τελικά ε, φαίνεται να μην λειτουργεί το σύστημα και με ποιον τρόπο, ποια είναι τα σφάλματα του. Και εγώ θα το πω ξεκάθαρα, το σύστημα λειτουργεί περισσότερες φορές μια χαρά. Όταν λοιπόν κάτι πάει στραβά, υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προσέγγιση όσον αφορά τους κινδύνους. Επικεντρωνόμαστε στους πολυάμεσους κινδύνους. Και ο κίνδυνος αξιολογείται στη βάση, σε μεγάλο βαθμό στη βάση ε, παραβιάσεις που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνει την υπόψη και το, το μέλλον. Επίσης, η έλλειψη ενδείξεων ε, χρησιμοποιείται και ως ένδειξη έλλειψης. Αυτό το λέω και εννοώντας ότι όταν δεν έχουμε ενδείξεις ε, για καταχρήσεις ε, θεωρείται ότι μάλλον δεν γίνονται. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το λογικό άλμα για να συνάγει κανείς από αυτό ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι ασφαλής απλά και μόνο επειδή δεν έχει κανείς ενδείξεις για το ότι έχουν υπάρξει παραβιάσεις ή καταχρήσεις. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου κράτη λένε ότι δεν έχω δει, ε, δει καταχρήσεις συγκεκριμένου εξοπλισμού στρατιωτικού. Αν και το ίδιο κράτος ενδεχομένως να έχει ε, προβεί σε κατάχρηση παρόμοιου εξοπλισμού. Αυτό ε, χρησιμοποιείται πολλές φορές ως δικαιολογία για την ε, τεκμηρίωση της ορθότητας μιας εξαγωγής. Όπως είπα, είναι δύσκολο. Το, είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε ε, σε ένα αποτέλεσμα. Αλλά η Αραβική Άνοιξη είναι ένα παράδειγμα όπου τα πράγματα πήγαν πολύ στραβά. Υπήρχε ένα βίο καθεστώς. Υπήρχαν για πολλά χρόνια εξαγωγές προς, προς αυτό το καθεστώς ή προς αυτά τα καθεστώτα και φαίνεται ότι αυτό συνέβη κιόλα ότι όταν κάτι πάει στραβά, πάει πολύ στραβά εάν τους έχεις προμηθεύσει, αν έχεις προμηθεύσει αυτά τα κράτη με όπλα. Και εδώ είχα μια συζήτηση με αξιωματούχο της ΚΟΑΡΜ και ε, με ρώτησε τι πιστεύαμε ότι θα συνέβαινε αν, όταν θα πέθαινε ο Καντάφη, ακόμη και αν πέθαινε από βαθιά γεράματα. Επίσης, το ότι τα τα κριτήρια αυτά θα πρέπει διαρκώς να υπηρετούν την ασφάλεια, τα οικονομικά συμφέροντα πάλι δεν ε, εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο. Επίσης, ε, σε άλλη συζήτησή μου με εξωματούχα του, της ε, ΚΟΑΡΜ μου είπε ότι πολλές φορές λάμβαναν αίτημα και αν δεν εγκρινόταν ε, οι ετούντες ζητούν, παρενέβαιναν σε υψηλότερο επίπεδο πολιτικής προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση. Μου υπόθηκε ότι αυτό πλέον αλλάζει και ότι η συζήτηση στο πολιτικό επίπεδο θα προηγείται της υποβολής αίτησης έκδοσης άδειας προκειμένου να μην ε, υπάρχει αυτού του είδους η πολιτική παρέμβαση προς τους αξιωματούχους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ε, μπορεί να βρεθούν και άλλες λύσεις. Και εγώ ε, δεν θέλω να πω ότι ο κλάδος έχει κάποια, είναι κακόβουλος. Ο κλάδος υπάρχει για τα συμφέροντά του προφανώς και θέλει να τα προωθήσει. Είναι οι κυβερνήσεις και η διακυβέρνηση του συστήματος που θα πρέπει να λαμβάνει τις, αποφάσεις, τις σωστές αποφάσεις. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα σύστημα που βασίζεται στα κριτήρια ε, λειτουργεί στις μεγάλες υποθέσεις. Αλλά όταν αρχίζει ε, αρχίζουν τα στρατηγικά και τα οικονομικά συμφέροντα να διονγκώνονται ε, και να γίνονται όλο και μεγαλύτερα, τότε αυτό το σύστημα που βασίζεται σε κριτήρια αρχίζει και υποφέρει. Και νομίζω ότι η ανάγκη τροποποίησης τους ε, είναι επιτακτική. Η Βόρεια Αφρική, η Αραβική Άνοιξη, η σχέση μας με τη Ρωσία, το καταδεικνύουν όλο αυτό. Και επίση υπάρχουν και ενδείξει απόκληση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκληση υποφέρει. Ε, λόγω των εξωτερικών πιέσεων ε, υπάρχει μια διαρκή στάση προς απόκληση αντί για σύγκληση. Υπάρχουν χώρες που θεωρούν ότι η αμυντική του βιομηχανία δεν συντελεί όσο σημαντική θα έπρεπε για την γενική τους οικονομική ε, ε, ευμερία. Uh, και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο ε, μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, έχω και μία άλλη ανησυχία, την ενσυνειδητότητα για αυτούς τους ε, νομικούς κανόνες, γιατί υπάρχει μία γνωσή τους. Άκουσα πολλές φορές πολιτικοί από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να λένε ότι αυτή η, χώρα δεν τελεί υπό ελμπάργκο, άρα μπορούμε να πουλήσουμε. Είναι νόμιμη η πώληση, αλλά δεν λειτουργεί έτσι η κοινή μας θέση. Ή η πώληση των Μιστράλ από τη Γαλλία στη Ρωσία. Από ό,τι γνωρίζω με την έκθεση του ΓΡΙΠ είδαμε καταρχήν πώς είχε η κατάσταση και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε γύρω από την πώληση. Και στη Γαλλία κανείς δεν αναφέρθηκε στα κριτήρια της κοινή θέσης. Δηλαδή το όλο θέμα ετέθη υπό διαφορετικούς όρους. Και η Ουκρανία ήταν αυτή που χρησιμοποίησε όρους της κοινή συμφωνίας. Αυτή είναι η μεγάλη ηρωνία, δεν προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ρωσία επίσης αναφέρθηκε στην κοινή ε, θέση όταν έγινε λόγος για πωλήσει από την Ουγγαρία στην Ουκρανία τάγκς ε, και εξοπλισμού. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την όλη κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο εμπροστοβαροί στην προσέγγισή μας. Ε, το είδαμε και με τη Γάζα και το Ισραήλ, όπου είδαμε ότι η διαδικασία διοδότησης είναι διαφορετική, εξαρτάται από το κράτος, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι υπάρχει μία πλημμυρίδα ανάλογα με το επίπεδο έντασης στη Γάζα. Δηλαδή οι όροι ε, συρρυκνούνται και διευρύνονται ξαφνικά. Μέσα σε μία δεκαετία ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Και θα δείτε περισσότερες, ε, περισσότερη σύραξη στη Γάζα. Δεν ξέρουμε πότε αλλά θα υπάρξει σύραξη. Και ίσως θα πρέπει να υπάρχει μία πιο ενιαία πολιτική εξαγωγών σε αυτή την περιοχή διαχρονικά. Υπάρχει επίσης και η έννοια της ε, ανάλυσης σε δύο στάδια. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε και από πλευράς ε, βιομηχανιών ή εταιριών ασφάλειας μέσα στα πλαίσια μιας αναλογιστικής προσέγγισης. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, πιο χρήσιμο, τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτή τη ε, διαδικασία διτής προσέγγισης, δηλαδή όταν ο κίνδυνος είναι χαμηλός, τότε η απόφαση είναι να εξαγάγουμε ακόμα κι αν οι συνέπειες αυτού του κινδύνου είναι υψηλές. Νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δύο ε, προσεγγίσεις στη διαδικασία αδειοδότησης. Επίσης θα ήταν σκόπιμο τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να βλέπουν το θέμα της διευκόλυνσης πιο λεπτομερός, και σε αυτή την περίπτωση η, συνθήκη πάει πιο μακριά από την κοινή θέση, γιατί η κοινή θέση ε, μιλά για διαδικασία πώλησης, ενώ η συνθήκη Άμστρεντ μιλά για διευκολύνσεις, δηλαδή μια ε, ευρύτερη εμβέλεια εφαρμογών. Δηλαδή δεν μιλάμε για το κατά πόσο υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς εξοπλίζουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό το βλέπουμε και με τη συνθήκη πώλησης ε, ή εμπορίας όπλων. Και το παράδειγμα των ε, κρατούμενων ίσως είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ίσως ο εξοπλισμός να μην χρησιμοποιείται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δημιουργεί τον τρόπο και τις προϋποθέσεις για το κράτος να δράσει υπό μία ορισμένη οπτική γωνία ως προς την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει ε, τρόπος και τόπος για νέα κριτήρια ή, ή διαφθορά για παράδειγμα, δηλαδή μπορώ εγώ να σας συντάξω ένα κριτήριο διαφοράς, το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο και να δούμε κατά πόσο, για να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένας κίνδυνος ε, σοβαρής διαφθοράς σε ένα κράτος και σε αυτή την περίπτωση δεν μεταφέρεται όπλα. Αυτό την χάνει επίκρισης γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε τη διαφθορά αλλά η ευρωπαϊκή κοινή προσέγγιση δεν βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, αλλά σε ανάλυση κινδύνου. Επίσης, ως προς τη διακυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έντονη γλώσσα, δηλαδή τις κατευθυντήριες γραμμές που ανέφερε ο προλαλής σας, και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα ισχύσει και όχι μόνο στις φτωχότερες χώρες αποδοχής η πώληση των όπλων. Υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα και ε, δημιουργεί μια μεγαλύτερη πρόκληση. Η πολιτική νομιμότητα, η υποστήριξη δεσποτισμού, τυραννίας, απολυταρχικών καθεστώτων και ούτω καθεξής, δηλαδή να πωλήσουμε όπλα σε ένα κράτος που γνωρίζουμε ότι είναι αυταρχικό ή θεωρείται αυταρχικό και του δίνουμε νομιμότητα και εμπιστοσύνη και αυτό υποσκάπτει τη δυνατότητα πολιτικών, πολιτικής διαμαρτυρίας, ειρηνικά από την αντιπολίτευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, πρέπει να μας απασχολήσει και μας οδηγεί σε ένα πιο πολιτικό πεδίο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των όπλων και σε τεχνικό επίπεδο. Και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν δεσμεύσεις σε πολιτικό επίπεδο Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα στο μέλλον και αυτό σχετίζεται με μια, ε, ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών άμυνας και παραγωγής για εγχώρια χρήση για να αντιμετωπίσουμε την ε, τρομοκρατία εύνης να δούμε τις συμμαχίες μιας χώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση επί του θέματος, αν και τώρα δεν υπάρχει τέτοια βούληση. Τώρα, στην περίπτωση της Ιεμένης, Κύριε Ίσπιξ, θα πρέπει να φτάσετε στα συμπεράσματά σας, γιατί θα έχουμε και δεύτερο γύρο. Άρα, για να αναφερθώ στην περίπτωση της Ιεμένης, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μεγάλη ε, εξάρτηση από τις πωλήσει σε αυτή την ε, περιοχή του κόσμου και πολλά ε, κράτη στην ουσία εγκύπτουν σε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά πέρα από την κοινή θέση. Έχετε την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας και της Σουηδίας την πώληση όπλων, όπου υπάρχει ένα μνημόνιο συνεννόησης. Δηλαδή υπήρχε μία ανταπόκριση του ευρύτερου ε, τομέα του εμπορίου στη Σουηδία που φοβήθηκε ότι εάν καταργηθεί το μνημόνιο συνεννόησης, αυτό θα είχε ευρύτερες επιπτώσεις στη ε, σουηδική βιομηχανία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ε, ισχύει πραγματικά αλλά έχει σημασία να δούμε κατά πόσο εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Δηλαδή, η οικονομική ευημερία βρίσκεται στα χέρια της πώληση όπλων προς αυταρχικά, καθαρά αυταρχικά καθεστώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάν Πι του αεροδιοστήματος και της άμυνας των, της Ένωσης της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ κυρίες και κύριοι για να αναφερθώ σε αυτό το θέμα του ελέγχου εξαγωγών όπλων εκ μέρους ε, της, ε, ε, του οργανισμού μας. Σήμερα θα αναφερθώ στο αμυντικό κομμάτι που καλύπτει ο οργανισμός μας να υπενθυμίσω ότι καλύπτουμε περίπου 3.000 εταιρείες, 50 άμεση ε, ε, συμμετοχή στο ESD και οι υπόλοιπες συμμετέχουν σε διάφορες ε, σε διάφορους οργανισμούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Πρώτον, για το θέμα των εξαγωγών και την αγορά εξοπλισμών, ε, όπως αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές, είναι διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα, από όλες τις υπόλοιπες αγορές. Είναι διαφορετική υπό την έννοια ότι οι αποφάσεις ε, για την χορήγηση αδειών είναι τμήμα της, ε, πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής της κάθε χώρας. Ειδικότερα όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεις συμμετέχουν άμεσα στι διαπραγματεύσεις και πάντοτε συμπεριλαμβάνουν ευρύτερα θέματα εθνικής ασφάλειας ε, και βασίζονται στους κυβερνητικού στόχου της κάθε χώρα τα ειδικά εθνικά συμφέροντα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική των κρατών μελών ε, ε, υπερισχύουν ε, του κέρδους για τις αγορές αυτές. Τα τελευταία, πέντε χρόνια, τα τελευταία χρόνια από το τέλος του ψυχρού πολέμου όλες οι κυβερνήσεις των κρατών που παράγουν όπλα τους ζητήθηκε να εξομαλύνουν κάπως την παραγωγή τους, να γίνουν κάπως πιο ε, ε, ιδιωτικού χαρακτήρα, να μην ε, δέχονται επιδοτήσεις, κάτι το οποίο τον κλάδων μας τον οδήγησε περισσότερο στις εξαγωγές. Αν δούμε το επίπεδο του προϋπολογισμού, βλέπουμε εθνικούς προϋπολογισμούς που συρρυκνώνονται, έχουμε δει όγκος, όγκο παραγωγών που μειώνεται και η μείωση του προϋπολογισμού είχε ως αποτέλεσμα ε, μια, ένα δύσκολο, μια δύσκολη πορεία για τις εξαγωγές μας, οι οποίες γίνονται όλο και πιο σημαντικές για, το, για τη βιομηχανία μας, για να μπορέσει να ε, επιβιώσει. Εμείς δεν μπορούμε να εξάγουμε παρά μόνο αν ε, δώσει άδεια για την κάθε εξαγωγή η κάθε κυβέρνηση είναι πολλά που διακυβεύονται. Η ανεξαρτησία της ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει για μεγαλύτερη τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία και αυτό πραγματικά είναι δύσκολο με τα λίγα εγχώρια ε, συμβόλαια, τα λίγα εγχώρια συμβάσεις που βλέπουμε σήμερα. Η κατάσταση λοιπόν ε, σημαίνει ότι πρέπει να επανέλθουμε στο βασικό ερώτημα, είναι μια πολιτική επιλογή την οποία πρέπει να συζητήσουμε. Η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει ένα επίπεδο στρατηγικής αυτονομίας και αν η απάντηση είναι ναι, σε ποιους τομείς θα ήταν αυτό, τι τεχνολογικές και βιομηχανικές υποδομές χρειαζόμαστε για να γίνει κάτι τέτοιο και τι θέλουμε να κάνουμε για τη διατήρηση των ε, υποδομών αυτών, τι σημασία θέλουμε να δώσουμε στις εξαγωγές. Τώρα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία και επειδή έχουμε δει πιέσει ε, στου εθνικού προπολογισμού ε, λιγότερα συστήματα ε, παράγονται για κάθε νέα γενεά οπλικών συστημάτων, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών. Είναι αναγκαιότητα πλέον, δεν είναι απλώς μια επιλογή. Αν όμως καταφέρουμε να διαχειριστούμε περισσότερη να επιφέρουμε περισσότερη συνεργασία, παρόλα αυτά οι εξαγωγές ε, θα εξακολουθούν να, παραμείνουν, να παραμένουν ζωτική σημασίας, με τρόπο όμως που πρέπει να είναι δυνατό να τον φέρουν τα κράτη-μέλη. Ε, πρέπει οι εταίροι να έχουν εμπιστοσύνη ότι κάποιο κράτος μέλος ε, δεν θα μπλοκάρει την εξαγωγή ανταλλακτικών σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, κάτι το οποίο θα επηρεάζει πολύ τις εξαγωγές μας και έχουμε δει παραδείγματα μιας τέτοιας κατάστασης. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, τότε η ευρωπαϊκή συνεργασία θα χαθεί και πολύ γρήγορα μάλιστα. Οπότε τα κράτη-μέλη είναι οι βασικοί εταίροι. Τα, τα κράτη-μέλη πρέπει να βρουν έναν τρόπο να εξασφαλίσουν ότι οι εσωτερικέ μεταφορέ ε, υπό ε, συστημάτων ε, πρέπει να συνεχίσουν και να είναι αντικείμενο ενός συστήματος συνεργασίας. Τώρα όσον αφορά την νομοθεσία, η εθνική νομοθεσία, ε, η οποία αντικατοπτρίζει τα κοινά, τις κοινέ αρχές της κοινής θέση του 2008 αλλά η εξαγωγή όπως αυτή διέπεται από τα συστήματα, από τα καθεστώτα εξαγωγής όπλων, ε, δυσκολεύει την κατάσταση, όπως δυσκολεύει και την κατάσταση ότι δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη μέλη των ιδίων πολυμελών οργανισμών, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα, ε, υπάρχουν διάφορες νομοθεσίες που πρέπει να, να ακολουθηθούν. Πρέπει να βρεθεί ένας διακανονισμός ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, ε, το έλυσαν αυτό το πρόβλημα από τα αεροσκάφη μέχρι τα πολεμικά πλοία, μέχρι τα ανταλλακτικά, μέχρι την τεχνολογία. Ε, μία από τις σημαντικότερες πτυχές για τον κλάδο ε, είναι η σαφήνεια και η προβλεψιμότητά του στα εθνικά συστήματα εξαγωγών όπλων αλλά και στους καταλόγους ελέγχων ε, που βρίσκονται πίσω από τα συστήματα αυτά. Αυτό είναι η σπονδυλική στήλη των διαφανών ελέγχων όπως επίσης και ε, του επιχειρηματικού προγραμματισμού. Αν λοιπόν ε, δούμε πώς έχουν τα πράγματα στη διεθνή σκηνή. Οι πέντε βασικοί προμηθευτές κατά το 2009 μέχρι το 2013 θα δείτε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν το 29% των παγκοσμίων εξαγωγών, Ρωσία 27%, μετά Γερμανία, Κίνα, ε, Γαλλία με 7, 6 και 5% αντιστοίχως. Πέντε, λοιπόν πρώτη εξαγωγής είναι το 75% της συνολικής εξαγωγής όπλων ε, ε, παγκοσμίως. Επομένως, κάποια κράτη-μέλη είναι πιο σημαντικά από άλλα, από απόψεως εξαγωγών ε, ή για τις ε, ευκαιρίες ε, στην αλυσίδα νηφοδιασμού ή ως πελάτες. Πολλές φορές οι πολυεθνικές δραστηριοποιούνται σε ε, παγκόσμιο ε, επίπεδο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε διεθνώς, δραστηριοριακά... και ζητούμε ε, συμμόρφωση με τα υψηλότερα κανονιστικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας. Ζητούμε, έχουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές βάσει του κώδικα δεοντολογίας για την αγορά και τις εξαγωγές όπλων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δεοντολογία και ακεραιότητα και είναι μεγάλη σημασία στρατηγικής αυτό και για το παρόν και για το μέλλον. Στο παγκοσμιούμενο περιβάλλον σήμερα πρέπει, πρέπει καθένας, κάθε χώρα να διαχειριστεί ε, την, ε, την επιβίωσή τους στις διεθνείς αγορές. Ε, εμείς μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας μας θέσαμε, διατυπώσαμε ένα έγγραφο δεοντολογίας, την επιμέλεια που πρέπει να δείχνουμε όταν, κάνουμε, όταν συνάπτουμε συμβάσεις με τρίτες χώρες και τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε διεθνή προγράμματα συμμόρφωσης και αυτό έγινε και μέσω του AST και με των εθνικών ενώσεων και οργανισμών σε πάνω από 4.000 εταιρείε σε όλη την Ευρώπη. Θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα ε, μαζί με το AIA, ε, τον, ε, τους Αμερικανούς ομολογούς μας, να έχουμε το IF bec δηλαδή μια ε, μια δεοντολογία που να μας ενώνει, ε, που να μας βρίσκει σύμφωνους και να επιτρέψει μια καλύτερη εξαγωγή όπλων σε Διεθνέ επίπεδο, όσον αφορά τώρα τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων από πλευρά ε, κλάδου και όπω το είπα, ότι, όπως είπα και προηγουμένω, η βασική προτεραιότητα είναι η συμμόρφωση με τα πρότυπά μα όπου γίνονται συναλλαγέ. Η οι δικές μας ε, οι, οι, οι διατάξεις της συνθήκης αυτέ, αυτής μερικές φορές πηγαίνουν πέρα από κάποια διεθνή μέσα που υπάρχουν. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια κενά που πρέπει να καλυφθούν. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει πρόοδος ε, ε, στο θέμα της ε, εκτροπής ε, όπλων ε, στο, στις παράνομες αγορές είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους ισότητας. Ποιος δηλαδή κερδίζει στο παιχνίδι αυτό. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία συμφωνεί λοιπόν με τη συνθήκη και τα μέτρα που περιλαμβάνει ε, και καλεί τα συμβαλόμενα μέρη να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις παράνομες δραστηριότητες. Πιστεύουμε ότι η συνθήκη θα ανεβάσει ψηλά τον πύχη σε παγκόσμιο επίπεδο και θέλουμε οι αντίστοιχες κυβερνήσεις μας να την επικυρώσουν και να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη συμμετοχή και την εφαρμογή ε, και από άλλες χώρες μέλη δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση το νόμιμο εμπόριο να υπονομευθεί από την εκτροπή όπλων σε παράνομες αγορές ή για χρήση σε δράσεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Επομένως η συνθήκη ε, θα ε, ισχύει και για χώρες στις οποίες ε, δεν υπάρχει σωστός έλεγχος των εξαγωγών όπλων. Μια καλή πρακτική θα έπρεπε να ενσωματώνει μια ανοιχτή κυβερνητική προσέγγιση για τους στόχου εφαρμογής της συνθήκης για το εμπόριο όπλων και πιστεύουμε ότι η αμυντική βιομηχανία πρέπει να ενημερώνεται για κάθε ε, αλλαγή στην νομοθεσία και να υπάρχει διαβούλευση μαζί της. Όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις ώστε να υπάρχει συμμόρφωση σε όλες τις ε, ε, δικαιοδοσίες οποίες ισχύει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει ένας πίνακας αξιολόγησης που ε, θα είναι πολύ σημαντικός κατά τη γνώμη μας και πολύ χρήσιμος παρά το γεγονός ότι γίνεται εφαρμογή της συνθήκης σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να είναι και συμβατή με την ε, ενωσιακή εσωτερική αγορά. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω για να σας δώσω μία σύνοψη της, της, του, της δικής μας, του δικού μα οργανισμού. Εμεί πιστεύουμε ότι είναι μία σημαντική αγορά η αγορά του εμπορίου όπλων ε, με τις συρρυκνούμενες δαπάνε ε, τα τελευταία 25 χρόνια. Οι εξαγωγέ έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές σημαντικές ε, και αυτό που διακυβεύεται είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Η ευρωπαϊκή συνεργασία εξαρτάται από τις εσωτερικές μεταφορές που δεν πρέπει να ε, ε, μπλοκάρονται μεταξύ κρατών μελών και σε παγκόσμιο επίπεδο το κανονιστικό πλαίσιο είναι πραγματικά πολύ πρόχειρο και δημιουργεί πολλές προκλήσεις για τη βιομηχανία μας. Ε, υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολύ υπάρχει πολλή νομοθεσία με την οποία πρέπει να συμμορφώνεται κανείς και αυτό που χρειαζόμαστε είναι σαφήνεια, ε, προβλεψιμότητα κοινώνου, ε, δεν μπορεί να αλλάξει κανείς τις αγορές του ή τους επιχειρηματικούς του εταίρους εν μια νυχτή. Είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Η επιχειρηματική ιδεοντολογια επίσης είναι βασική προτεραιότητά μας και θα παραμείνει. Ε, υποστηρίζουμε τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων που αποτελεί πραγματικά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ανοίγει ο κατάλογος ομιλητών για να υποβληθούν ερωτήματα και να δοθούν και απαντήσεις, αν έχουμε χρόνο βέβαια. Πρώτος ομιλητής είναι ο εισηγητής της Επιτροπής ε, ΣΕΝΤΕ, η εισηγήτρια η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω και πάλι σου ειδικά. Και γι' αυτό περιμένω να βάλουν όλοι τα ακουστικά του. Ο Γιάνν βέβαια με καταλαβαίνει έτσι κι αλλιώς. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν, αλλά ε, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ο Ρόι το ανέφερε λίγο. Ε, θα πρέπει δηλαδή να ε, εξετάζεται και η κατάσταση στην χώρα παραλήπτη. Υπάρχουν και ορισμένοι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει κανείς να ελέγχει για ποιον σκοπό προορίζονται αυτά τα όπλα και μπορεί κανείς να ναι ή όχι στη βάση αυτού του ελέγχου. Πρέπει δηλαδή να εξετάζεται και η κατάσταση στη χώρα παραλείπτει. Όχι μόνο όμως ε, ε, ο σκοπός χρήσης των όπλων. Στην ε, Σουηδία υπάρχει μια, ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητείται και όπου προβλέπεται ότι θα πρέπει να εξετάζεται αν η χώρα παραλήπτης είναι δημοκρατία ή αν πρόκειται για αυταρχικό καθεστώς ώστε να διευρύνεται και η βάση στην οποία, επί της οποίας αξιολογείται ε, μια απόφαση περί εξαγωγής ή όχι. Πρόκειται δηλαδή και για μια πολιτική απόφαση. Ποιες χώρες είναι αποδεκτές και ποιες όχι. Άρα ε, δεν μπορεί μοναδικό κριτήριο να είναι ο σκοπός χρήσης. Σκεφτείτε τη Σαουδική Αραβία. 50% του πληθυσμού δεν έχει καθόλου δικαιώματα. Δεν είναι αυτό ένα κριτήριο το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται και αυτό υπόψη. Υπάρχει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο που συζητείται στην Σουηδία που ε, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία και από αυτή την άποψη επηρεάζει και τους ε, ενδοευρωπαϊκούς, τις ενδοευρωπαϊκές ε, εξαγωγές, μεταφορές. για τη Σουηδία διαγράφεται, διαγράφονται πολλές δυσκολίες αν υπερψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο στην συνεργασία της με άλλες χώρες. Άρα χρειάζεται πολιτική σαφήνεια και ε, ενδεχομένως θα, θα μπορούσε και στην κοινή θέση να αναθεωρηθεί αυτή η βάση επί της οποίας λαμβάνεται η απόφαση για πώληση όπλων ή όχι. Επίσης, ε, αναφέρθηκε το ζήτημα της αγοράς. Ε, ο κλάδος ε, και των αγορών. Ο κλάδος ε, καταβάλει μακροχρόνιες προσπάθειες προκειμένου να ανοιχτεί συγκεκριμένε αγορές. Για παράδειγμα, καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να ανοιχτούμε στη Μέση Ανατολή, όπου ε, όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν δραματικές εξελίξεις και πολλές φορές τα ίδια τα όπλα που εμείς έχουμε πουλήσει στις χώρες αυτές λόγω της, αλλα... της αλλαγής της κατάστασης μπορεί να στραφούν και εναντίον μας. Δεν είναι τα πράγματα στην Μέση Ανατολή όπως ήταν το 2008 όταν καταλήξαμε στην κοινή θέση. Η κατάσταση έχει αλλάξει και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη εμείς εδώ στην Ευρώπη. Η κατάσταση ε, δεν μπορούμε διαρκώς μόνο να παραπέμπουμε στο γεγονός ότι δημιουργήθηκαν 8.000 θέσεις εργασίας στην αμυντική βιομηχανία, πρέπει να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο και για ποιον σκοπό έχουμε την αμυντική βιομηχανία. Και ο λόγος, ο σκοπός, ε, κατά τη γνώμη μου, είναι ε, να μπορούμε να αμυνθούμε σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ευρώπης. Φυσικά, μια αλλαγή της κοινή θέση ενδεχομένως να επηρεάσει και την αμυντική βιομηχανία, αλλά παρόλα αυτά επιμένω ότι θα πρέπει την ε, συνολική κατάσταση να την ε, αξιολογούμε και να την κρίνουμε με βάση την, τρέχουσα ε, ε, κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια. Επίσης, όσον αφορά τα εμπορεύματα διπλής χρήσης, ε, στον κατάλογο υπάρχουν πάρα πολλά ε, αγαθά τα οποία δεν αναφέρονται. Παρόλα αυτά όμως θα μπορούσαν αυτά τα αγαθά στα οποία αναφέρομαι να χρησιμοποιηθούν κατά του πληθυσμού, κατά των λαών. Άρα πρέπει να αναθεωρηθεί και ο κατάλογος. Και ένα άλλο σημείο το οποίο δεν αναφέρθηκε. Εξαρτιόμαστε όλο και πιο πολύ από τις εξαγωγές Υπάρχει όμως και η τεχνολογία που αναπτύσσει η βιομηχανία. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και την βιωσιμότητα, τη βιωσιμότητα μάλλον και αυτού του κλάδου. Ευχαριστώ ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις παρουσιάσεις. Αρχικά να πω ότι συμφωνώ σε αρκετά σημεία με την συνάδελφο Βαλέρο, ιδιαίτερα συμφωνώ ότι κατά κύριο λόγο θα πρέπει ε, να υπάρχει αμυντική βιομηχανία με κύριο σκοπό να μπορούμε να αμυνθούμε σε περίπτωση κρίσης. Και από αυτή την άποψη το επιχείρημα περί δημιουργίας θέσεων απασχόλησης είναι έολο, γιατί με αυτό το επιχείρημα θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει οποιαδήποτε εξαγωγή. Η βιομηχανία και οι εμπειρογνώμονες που διαθέτουμε είναι και το παράπλευρο ε, κέρδος, πλεονέκτημα που έχουμε, από το γεγονός όμως ε, που απορρέει από μια συγκεκριμένη ανάλυση περί απειλών την οποία κάνουμε. Δηλαδή, λέμε ότι πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αμυνθούμε σε περίπτωση πολέμου, γι' αυτό καλώς έχουμε αμυντική βιομηχανία και γι' αυτό το λόγο ε, θεωρώ και εγώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο στρατηγικής αυτονομίας. Δηλαδή, με ίδια μέσα θα πρέπει να μπορούμε να ε, υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και τις χώρες μας. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει για τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Από αυτή την άποψη το, το ΝΑΤΟ είναι αναντικατάστατο. Απλά μιλώ για τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εδώ στη γειτονιά μας. Θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, στη γειτονιά μας δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, αυτόνομοι. Ε, για να μην υπάρχει και ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε κάποιο βέτο από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζω το αίτημα περισαφήνειας και προβλεψιμότητας ε, της, ε, του αμυντικού, της αμυντικής βιομηχανίας, του κλάδου. Χρειάζονται όλα αυτά ακριβώς γιατί μιλούμε για επενδύσεις, ε, επενδύσεις και σε ανθρώπινο δυναμικό και στην έρευνα και γι' αυτόν τον λόγο η ε, πολιτική θα πρέπει να ε, αποφύγουμε απρόβλεπτες αλλαγές. Νομίζω ότι μία από τις απαντήσεις που δεν δόθηκαν σε σύνοδο των Υπουργών Άμυνας είναι το ζήτημα της ασφάλειας τροφοδοσίας που μάλιστα είχε ανατεθεί ως καθήκον από, το προηγούμενο, από την προηγούμενη σύνοδο στην Κομισιόν να υποβάλει δηλαδή πρόταση. Δυστυχώς τέτοια πρόταση δεν υπήρξε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η επιδίωξη είναι συμβατή με την τροποποίηση των εθνικών νομοθεσιών όλα εκείνα τα στοιχεία που ε, οδηγούν σε κοινέ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν δηλαδή αποφασίζουμε να κάνουμε κοινέ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας θα πρέπει να εξασφαλίζεται να ικανοποιούνται τα, τα αιτήματα που υποβάλλονται από κράτη-μέλη. Θα ήταν αντίφαση να λαμβάνονται ομόφωνες αποφάσει και στη συνέχεια να μην υλοποιούνται. Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, πιστεύω ότι πέρα από την κοινή θέση θα πρέπει να πραγματοποιείται και μια κατά περίπτωση ανάλυση. Αν για παράδειγμα σε τρίτες χώρες αλλάξουν οι συνθήκες κάποια στιγμή, θεωρώ ότι μπορεί κανείς, θα μπορεί κανείς να ε, εξάγει όπλα και σε αυταρχικά καθεστώτα ε, αν για παράδειγμα το καθεστώς αυτός πρόκειται να καταπολεμήσει, να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό κράτος. Υπάρχει η κατάσταση όπου μία ε, μη ε, κρατική οντότητα ε, προκαλεί εξαθλίωση. Αν λοιπόν δεν είσαι εσύ έτοιμος να παρέμβεις, τότε θα πρέπει να μπορείς τουλάχιστον να συνυπολογίζεις και άλλους ε, παράγοντες. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο ευελιξίας όσον αφορά την κοινή θέση, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα, να διατηρούμε τη δυνατότητα ε, να αντιδρούμε ε, στις ξεκαταστάσεις που ενδεχομένως να αλλάζουν. Ευχαριστώ κύριο Σκάν. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ και εγώ τους τρεις ομιλητές για το ότι φώτισαν διάφορες διαστάσεις. You talked about 20... Είπατε ότι 20 χώρες έχουν υπογράψει και απομένουν δύο. Ποιες είναι οι δύο. Επίσης μιλήσατε για το Ηνωμένο Βασίλειο που έδωσε άδειε στα πλαίσια της ε, ε, Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας. Πώς έχει η διαδικασία αυτής της αδειοδότησης. Το άλλο που θα ήθελα να ε, ακούσω είναι οι απόψεις των τριών ομιλητών ως προς όλο αυτό το θέμα που σχετίζεται με τη διαφθορά και την πώληση όπλων. Βεβαίως η διαφθορά δεν είναι αποδεκτή, αλλά με ορισμένες ε, χώρες του τρίτου κόσμου είναι σαν να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιες είναι οι αντικσότητες το θέμα του χρέους που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές οι χώρες, καθώς και ε, το, το θέμα της καταπίεσης προς αυτές τις χώρες, γιατί η πολιτική αρχή δημιουργεί αστάθεια και πολλές φορές αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία πολιτική αντιμετώπιση του μεγαλύτερου κύματος προσφύγων μέχρι σήμερα. Και το θέμα της Μέσης Ανατολής βέβαια. Μιλάμε για εκατομμύρια πολλών δις προς τη Μέση Ανατολή. Και είπαμε ότι θα πρέπει οι βιομηχανίες μας να επιβιώσουν. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά από ορισμένα κράτη, γιατί πολλοί θέλουν να βγάλουν δισεκατομμύρια από την πώληση όπλων, αλλά αντιστρέφονται στους ανθρώπους, δηλαδή υποστηρίζουν δικτατορικά καθεστώτα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και αυτό το, το στοιχείο του, του διπλού μέτρου. Ε, κάτι άλλο που απορρέει από την τελευταία μου δήλωση αφορά τις τρέχουσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Πώς σχετίζεται με το εμπόριό μας, με την τακτική μας πώληση όπλων ανά τον κόσμο. Δηλαδή μας ενδιαφέρει το ε, βραχυπρόθεσμο χρέος και μόνο. Τη στιγμή που μιλάμε για ε, βραχυπρόθεσμο κόστος με, μακροχρόνιο, με ένα μακροχρόνιο ε, εύρος δυστυχιών. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να δούμε και τις χώρες οι οποίες εισάγουν αυτά τα αμυντικά όπλα. Εδώ υπάρχουν και η Ινδία και το Πακιστάν. Γνωρίζουμε ότι είναι μια περιοχή σειράξεων. Είχαμε τρεις πολέμους και βεβαίως υπάρχει και ο κίνδυνος των πυρηνικών. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε και να εξοπλίζουμε αυτές τις χώρες όλο ένα και περισσότερο γιατί αυτό καθε αυτό θα μπορούσε να είναι επιζήμιο στην παγκόσμια ειρήνη. Ο Μάρεκ Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, όλους τους πάνελιστ για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και input. Η τα κριτήρια ως προς τις εξαγωγές όπλων θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Θα πρέπει να έχουμε πιο, μια πιο ολιστική ε, προσέγγιση στο θέμα. Το θέμα της εθνικής ασφάλειας αφορά την προστασία των ανθρώπων από ενδυνάμει απειλές και πραγματικές απειλές. Ίσως και αυτό θα πρέπει να είναι ε, πρόκριμα των δράσεών μας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δούμε συγκεκριμένες χώρες, την κυβέρνησή τους και τη θέση τους ως προς τη συλλογική ασφάλεια. Και επίσης δεν θα πρέπει να τιμούμε περισσότερο και τη δική μας θέση. Νομίζω ότι όλες, μας, όλες οι χώρες θα πρέπει να, να τιμήσουν τη θέση των ε, χωρών του Νότου σε σχέση με τη Μεσόγειο. Είτε αυτό αφορά την Πολωνία είτε τις Βαλτικές χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει η ίδια προσέγγιση ως προς το Νότο. Τα πλοία Μιστράλ που μετέφεραν Μιστράλ δεν θα έπρεπε να έχουν μεταβεί στη Ρωσία. Είναι μια χώρα η οποία ε, προωθεί την εμπόλεμη σύραξη στην Ουκρανία. Γι' αυτό και αυτή η απόφαση δεν έπρεπε να ληφθεί ποτέ. Επειδή θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σωστό επιμερισμό βαρών ως προς τις θέσεις μας, γιατί πολλοί προβάλλουν δικαίωμα αρνησικυρίας αλλά βέβαια είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και η εθνική ασφάλεια είναι ένα θέμα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όσοι εξάγουν όπλα στη Ρωσία μας λένε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία ε, μεταβαίνει στη δημοκρατία. Δείτε όμως την κατάσταση στο Ιράν και την κυβέρνησή του. Νομίζω ότι δεν πρέπει να εξάγουμε ούτε στο Ιράν, αλλά ούτε και στη Ρωσία με βάση τη θέση τους. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μία ψυχρό ανάλυση των κριτηρίων εξαγωγών και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα τη, μέσω της συνεργασίας. Επίσης, το διεθνές εμπόριο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ε, πολιτικής μας ασφάλειας. Αυτά που είπα για τη Ρωσία έχουν σημασία και για ιστορικούς λόγους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε ορισμένες αποφάσεις. Έχουμε τον τρομακτικό πόλεμο της Ουκρανίας και αυτό άνοιξε τα μάτια του κόσμου. Όμως, εάν ε, προβάλλουμε μία πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Έτσι θα εμβαθύνουμε τη συνεργασία που προωθούμε και έτσι θα μπορούσαμε να ξαναδούμε τα κριτήρια των εξαγωγών όπλων ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής μας άμυνας και ασφάλειας, γιατί είναι μια πολιτική η οποία συμπίπτει και με τα συμφέροντα των κρατών μελών προς την ασφάλεια. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Με πολλές από τις θέσεις που ακούστηκαν συμφωνώ. Να ξεκινήσω από το επιχείρημα με τη δημιουργία, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και μελέτες που αποδεικνύουν ότι η σημασία της αμυντικής βιομηχανίας για την απασχόληση είναι πολύ μικρότερη από ότι πολλές φορές ε, θεωρείται ως δεδομένο. Ένα δολάριο, για παράδειγμα, στον κοινωνικό τομέα ε, δημιουργεί τριπλάσιες θέσει εργασία, από ότι ένα δολάριο που επενδύεται στην αμυντική βιομηχανία. Και εγώ συνεργάζομαι και με οργανώσεις στην ε, Γερμανία που έχουν ως σκοπό του τον αφοπλισμό και γνωρίζουν ε, ότι πολλοί από τους εργαζόμενους μάλιστα τη αμυντική βιομηχανίας θα ήθελαν να εργάζονται σε άλλους κλάδους αν είχαν τη δυνατότητα. Τώρα, συζητούμε τα κριτήρια και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κριτήρια. Πάντως, θεωρώ ωστόσο ότι είναι σημαντικότερο ε, η εφαρμογή, ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων. Ο, τα κριτήρια, όπως είναι διατυπωμένα αυτή τη στιγμή, επιτρέπουν τόσες πολλές παραβιάσεις και παραβάσεις που για μένα κοινωνιολογικά μια τροποποίηση των ε, κριτηρίων φαίνεται να είναι σημαντική, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να επιφέρουν πρακτικά αποτελέσματα αυτές οι αλλαγές. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να συζητήσουμε για τις δυνατότητες εφαρμογής αυτών των κριτηρίων, να συζητήσουμε ποια κενά ε, υπάρχουν στους ελέγχους ε, όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων, πώς μπορούν να καλυφθούν τα κενά αυτά και θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε τι θα κάνουμε σε περιπτώσεις παραβάσεων. Έχουμε συζητήσει και για κυρώσεις. Κάτι που βεβαίως μπορεί να πλήξει σε έναν μικρό βαθμό τουλάχιστον και τα κέρδη της αμυντικής ε, βιομηχανίας. Ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση πλέον δεν θα αξίζει και τον κόπο να ε, εξάγει κανείς αν έχει να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Να προσθέσω και ένα κριτήριο το οποίο δεν συζητήθηκε, το κριτήριο 8. Εκεί όπου γίνεται λόγος για το ότι θα πρέπει να εξετάζονται και οι χώρες παραλήπτες. Δεν θα πρέπει να εξετάζονται μόνο τα, οι διαστάσεις ασφάλειας, οι πτυχές ασφάλειας. Το κριτήριο λέει ότι θα πρέπει να ίζονται και τα αναπτυξιακά συμφέροντα του κράτους παραλήπτη. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να γίνονται εξαγωγές αν δεν έχουν οι χώρες παραλήπτες την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αυτά τα ε, όπλα. Όσον αφορά την, ε, τις μεταπολίσεις, ε, θεωρώ ότι και, αυτές, και αυτό είναι ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί. Επίσης, αναφέρεται συχνά ότι υπάρχει μια απόκληση όσον αφορά τα συμφέροντα των επιμέρους κρατών μελών. Συμφωνώ από πολλές απόψεις, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και το εξής. Δεν υπάρχει μόνο μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν αντιθέσεις και εντός της κάθε χώρας ξεχωριστά. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι ε, πολλοί κοινωνικοί κύκλοι, πολλά κοινωνικά στρώματα θεωρούν ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των εξαγωγών και ταυτόχρονα οι πολιτικοί εκπρόσωποι κινούνται σε μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης, αναφέρθηκε, ε, αναφέρθηκαν τα συμφέροντα της Ουκρανίας ε, σε σχέση με τη Ρωσία και εκεί πάντοτε συμφωνούμε. Υπάρχει συνένεση. Τι γίνεται όμως με τη Σαουδική Αραβία. Στο, στην περίπτωση αυτή η Άγγελα Μέρκελ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι η Σαουδική Αραβία είναι στρατηγικός εταίρος της Γερμανίας και γι' αυτό το λόγο εμείς ό,τι και να γίνεται στη χώρα αυτή θα κάνουμε εξαγωγές. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις Αν όμως δεν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούμε να καθόμαστε να μιλάμε τώρα για θέσει από απασχόληση κτλ. κτλ. Σε κάθε περίπτωση εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι θα πρέπει μια κοινωνία να συζητά ποιο είναι το ηθικό τίμημα που καλείται να πληρώσει για την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων. Ποια είναι η ηθική διάσταση, ποιο είναι το ηθικό τμήμα που είναι πρόθυμες οι κοινωνίες να πληρώσουν. Ευχαριστώ κύριο Σκέζα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί σήμερα το πρωί επιτελέστηκε μια πολύ θετική εργασία γιατί με τον πρεσβευτή Ποπόφσκι μιλήσαμε για την ενίσχυση της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Υπήρου μας. Και ασχοληθήκαμε με επιμέρους θέματα, πώς, ε, τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας μέσα στα πλαίσια και των ε, δημοσιονομικών ε, ενισχύσεων. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων και πώς να χρηματοδοτήσουμε τις 3.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να ενισχύσουμε και την ε, Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Ασφάλειας. Το πραγματικό όμως πρόβλημα είναι πώς να εποπτεύσουμε αυτόν τον τομέα σε σχέση με ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Το τωρινό πάνελ έχει άμεση σχέση με την προγενέστερη συζήτηση, δηλαδή μας ενδιαφέρει μια ενισχυμένη πολιτική ασφάλειας και βεβαίως και οι κατάλληλοι εξοπλισμοί. Πώς όμως μπορούμε εμείς να εξοπλίσουμε άλλους προκαλώντας ε, και προωθώντας έφλεκτες καταστάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Νότον, πώς μπορούμε να υποπτεύσουμε εμείς καλύτερα το θέμα των εξαγωγών. τα όπλα ε, πολλούνται με βάση ένα συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό τίτλο, αλλά βρίσκονται στα χέρια τρομοκρατών στη συνέχεια. Πόσο μπορούμε ε, αυτά τα όπλα τα οποία έχουν εξαχθεί νόμιμα και πολιθεί νόμιμα να μην μεταφέρονται σε χέρια τρομοκρατών. Μία άλλη έχει ως εξής πώς ε, θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε σε χώρες ε, το ενιαίο πλαίσιο εξαγωγών, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε αυτή την εργασία εποπτείας και ελέγχου στην όλη πολιτική εξαγωγών και εμπορίας όπλων. Ευχαριστώ. Κράσνοντάμσκι. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι κάπως διαφορετική. Θα ήθελα να σταθώ στην κατάσταση της Ευρώπης και να ρωτήσω τους, κυρίους ή σκέφτονται ως προς τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών, μελών και ευρωπαϊκών βιομηχανιών μέσα στην Ευρώπη. Πώς αυτές οι επιχειρήσεις ή χώρες συνεργάζονται για να υπεκφύγουν του ελέγχου εμπορίας ε, όπλων. Και εδώ λαμβάνω υπόψη την συγχώνευση της KMW και μίας αντίστοιχης γαλλικής επιχείρησης. Από ό,τι κατάλαβα, στόχος της συγχώνευσης ήταν να υπεκφύγουν την νομοθεσία εξαγωγής όπλων από τη Γερμανία. Κάτι τέτοιο συμβαίνει συχνά. Αυτό είναι ο τρόπος για να αποφύγει κανείς ή να υπεκφύγει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και μέσω συγχωνεύσεων. Ο εκπρόσωπος της S5 από το Bundestag, υπεύθυνο για θέματα ασφαλείας και άμυνας, μίλησε για το γεγονός ότι δεν πρέπει να πολλούνται τάγκς στη Γαλλία Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η δήλωση. Δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να αποτρέψει την πώληση όπλων σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για κοινή πολιτική όταν δεν προβαίνουμε σε αλληλοπολίσεις, μεταξύ μας δηλαδή. Άρα τι σκεφτόσαστε σε σχέση με την αποφυγή κανόνων, δηλαδή διευθετήσεις που υποσκάπτουν τους ίδιους τους κανόνες και δεύτερον, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών καθαρά συμφερόντων, ποια θα μπορούσε να είναι τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Να πω και χωρισμένα πράγματα για αυτές τις παρουσιάσεις. Θα ήθελα να αρχίσω καταρχάς με μία ερώτηση προς τον κύριο Λοτών. Υπάρχει μία συζήτηση για την ενδεχόμενη ανάγκη αλλαγής ε, του καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών όπλων. Ποια είναι η άποψή σας και ποια είναι η δική σας αξιολόγηση για το πού βρίσκεται αυτή η συζήτηση, τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ του παγκοσμίου και του ευρωπαϊκού καθεστώτος ελέγχου. Και θα ήθελα επίσης ε, να κάνω μια ερώτηση για τα, ερώτη... για τα όσα μας είπε ο κύριος Σπίστερ. Καταρχάς, Όταν μιλάμε για την κοινή θέση για τις εξαγωγές Μιστράλ ε, στη Ρωσία και για την ε, ενδεχόμενη εξαγωγή όπλων ε, στην Ουκρανία, νομίζω ότι κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος σε σχέση με την έγκριση των βασικών κριτηρίων. Το, το να το επαναλαμβάνουμε δηλαδή εδώ, γιατί όσον αφορά στη Ρωσία, για πολλά χρόνια είχαμε να κάνουμε με ένα επιθετικό κράτος. Για πολλά χρόνια νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ σιωπηλοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τώρα την πώληση Μιστράλ, δεν ήταν μόνο η Ουκρανία, ήταν η Πολωνία, ήταν και οι Βαλτικές χώρες, κράτη-μέλη της Ένωσης, ε, που ε, το είχαν ε, ε, πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα Μιστράλ, ξέρετε ότι είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα και μεταφορά τεχνογνωσίας, πολύ εξελιγμένης τεχνογνωσίας και δεν μιλάμε Δεν μιλάμε μόνο για στρατιωτικά, για πολεμικά πλοία, για πολύ περισσότερα μιλάμε. Και εμείς παραμένουμε σιωπηλοί, δεν λέμε τίποτα. Και όταν μιλάμε για, για τα κριτήρια και για την αναγκαιότητα έγκρισης ε, ε, οικουμενικών κριτηρίων, συμφωνώ ότι πρέπει να σκεφτούμε τα ε, ολοκληρωτικά καθεστώτα, αλλά πρώτα πρέπει να σκεφτούμε τα επιθετικά κράτη, και να προσπαθήσουμε να προλάβουμε την ε, πώληση ε, όπλων σε επιθετικά κράτη και δεν είναι δυνατόν ε, τη Ρωσία και την Ουκρανία να τις θέτουμε στην ίδια βάση και νομίζω ότι η κοινή θέση δεν είναι παρκής στην αξιολόγησή της των δύο αυτών περιπτώσεων. Όταν μιλούμε και κατά την άποψή μου η παρουσίαση του ε, Γιάνν Πι με έκανε να σκεφτώ πολλά πράγματα. Ε, συμφωνώ μαζί σας ότι ε, η αμυντική βιομηχανία και οι αμυντικές αγορές είναι πολιτικές αγορές. Όταν μιλήσατε για τη σημασία της διατήρησης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, αυτό εννοεί, με αυτό εννοείται ότι θέλουμε να είμαστε πολιτικά αυτόνομοι και επομένως πρέπει να σκεφτούμε να έχουμε μια κοινή θεώρηση του ωφέλους, των ε, ευκαιριών αλλά και των απειλών. Αυτό είναι το βασικότερο. Το πρώτο κριτήριο για την ανάληψη δράσης σε πολιτικό επίπεδο από κοινού και βέβαια όταν ε, θέλουμε να είμαστε στρατηγικά αυτόνομοι και έτσι να ε, ενεργούμε, πρέπει να σκεφτούμε και τους λόγους ύπαρξης των εθνικών στρατηγικών ε, προγραμμάτων, ε, γιατί από πολιτικής απόψεως είναι μια θεώρηση της εξωτερικής πολιτικής τους και της θεώρησης τους ε, για την πιθανή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το να κυριαρχεί η άποψη και μας δώσατε και συγκεκριμένες στατιστικές ε, οι οποίες είναι πολύ ουδέτερες, δηλαδή πόσο είναι κυρίαρχες αυτές ε, οι ε, χώρες, η Γερμανία και η Γαλλία στην αμυντική βιομηχανία, το να υπερισχύουν σε αυτό σημαίνει ότι περισχύουν και στην εξωτερική, ε, ε, ότι υπερισχύει και η θέση τους περί εξωτερικής πολιτικής είναι απλά τα πράγματα. Και το λέω αυτό ότι ίσως θα ε, γιατί πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξουν και επιπλέον κριτήρια για να αντιμετωπιστεί αυτό. Και το ερώτημα μου, το ερώτημα μου προς τον κύριο Ισμπίστερ, όταν παραθέτουμε παραδείγματα, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτά είναι πολιτικά παραδείγματα και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε να, να τηρούμε κάποιες ισορροπίες όταν παραθέτουμε τα παραδείγματα αυτά. Λωτό, Ισμπίστερ και μετά πι. Ευχαριστώ Καταρχάς, το εύκολο ερώτημα. Τα δύο κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ε, υπογράψει τη συνθήκη είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Μόνο αυτές δεν την έχουν επικυρώσει, ε, αλλά είναι ζήτημα μηνών. Θα ήθελα να σας πω για την ευρύτερη σύγκληση, το γνωρίζετε, η άποψη του Συμβουλίου είναι η εξής, ότι δεν θα παραβιαστούν οι κανόνες και η προσέγγιση, όπως γνωρίζετε, που έχει συμφωνηθεί από το 2012 δεν είναι η παραβίαση των κανόνων, αλλά η καλύτερη εφαρμογή τους. Επομένως υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποια μέσα στην κοινή θέση για την υποστήριξη της σύγκλησης και πρέπει, και αυτή είναι η προσέγγισή μας, να τα εφαρμόσουμε περισσότερο, πιο σωστά, με πιο επικοδομητικό και εφευρετικό τρόπο, ε, ε, το, δεν, δεν είναι ρεαλιστικό να σκεφτόμαστε βέβαια ότι μόνο αυτό ε, θα υποστηρίξει την σύγκληση. Είναι κάτι το οποίο παραμένει να το διαπιστώσουμε κατά τα επόμενα ε, χρόνια. Τώρα το ερώτημά σας ε, που αφορούσε την ε, ολοκλήρωση της αναθεώρησης και πότε θα είναι η επόμενη θα είναι το 2018, 10 χρόνια μετά την έγκριση της κοινή θέσης και τότε θα έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε όλες αυτές, ε, όλα αυτά τα, όλες αυτές τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουμε για την εφαρμογή. Μετά υπήρξε ένα ερώτημα όσον αφορά την, ε, ε, το ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την κατάχρηση της προμήθειας όπλων και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, αυτή η κακή χρήση της εξαγωγής όπλων, στο, στο κατά πόσο μπορούν δημοκρατικά να παραδοθούν αυτά τα τα όπλα. Είναι γεγονός. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί. Από την άλλη όμως, δουλεύει και αντιστρόφως. Όταν είναι κανείς ε, μια κυβέρνηση και έχει μια προμήθεια για μαχητικά αεροσκάφη που έχουν ένα κύκλο ζωής 30-40 χρόνια, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κίνητρο να μην ε, διαφωνήσεις ε, με τον προμηθευτή σου γιατί δεν θέλεις να βρεθεί σε μια κατάσταση στην οποία έχεις 15 ε, εκατομμυρίων δολαρίων αεροσκάφος στο έδαφος γιατί δεν υπάρχει το τάδε ανταλλακτικό που χρειάζεσαι γιατί έχει τσακωθεί με τον προμηθευτή. Λοιπόν, πρέπει να το δείτε και αυτό, να δείτε και την οπτική αυτή γωνία ότι για ραντάρ, για, ε, ε, για τάγκς, ε, για όπλα τα οποία έχουν κύκλο ζωής 50 χρόνια για παράδειγμα. Καλή είναι η προμήθεια, αλλά δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν δεν, δεν είναι δυνατόν να είμαστε βέβαιοι ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες ασφαλείας που υπήρχαν όταν συνήφθη η σύμβαση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ναι, πολύ καλές είναι οι εταιρείες ως προς την παράδοση των ε, ε, προϊόντων, αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρά τα κριτήρια για την τελική χρήση. Πρέπει να γίνεται επαλήθευση και επανέλεγχο συνεχώς. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι έχει κανείς ε, ε, εξασφαλίσει ότι πληρούνται όλες ε, οι προϋποθέσεις και πρέπει ως πελάτης να ξέρεις ότι για παράδειγμα αυτά που έχει παραγγείλει θα μείνουν στην αποθήκη του Υπουργείου Άμυνας και ότι δεν θα προωθηθούν κάπου αλλού με κάποιο σκοτεινό τρόπο. Προφανώς όσον αφορά τις άδειε, κάποιες από αυτές μπορεί να είναι αμφισβητήσιμες, αλλά τελικά έχουν κάποιους κανόνες και κάποιες προϋποθέσεις, κάποιους όρους από πίσω τους, που μπορούν να προσαρμοστούν, να μετριαστούν με κάποιο τρόπο, ώστε ακόμη περισσότερο να εξασφαλίζουν την κακή χρήση, την ενδεχόμενη κακή χρήση, ώστε να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη. Όσον αφορά τώρα την, το τι γίνεται μετά τη χορήγηση της άδειας, ότι πρέπει κανείς να είναι έτοιμος για μία βίαιη αλλαγή των συνθήκων και να πει κανείς ότι ναι, αυτή η προμήθεια δεν είναι δυνατόν να γίνει πια ε, όλα τα κρατημέλη μπορούν, δεδομένης κατάστασης με το Ισλαμικό κράτος, ε, έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τις ε, αδειές τους, ε, μπορούν να τις αναστείλουν και οι πελάτες μπορούν να μπλοκάρουν στα σύνορα το εμπόρευμα υπάρχουν κάποιες αν υπάρχουν άδειε οι οποίε ισχύουν ακόμα, υπάρχει το τελευταίο, η τελευταία δυνατότητα να ε, μπλοκαριστούν αυτά τα ε, προϊόντα, αυτά τα εμπορεύματα ε, στα σύνορα, λέγοντας ότι για παράδειγμα, ξέρετε, έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει συνθήκες και η άδεια δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται πλέον, γιατί η άδεια πρέπει να ανασταλεί ή γιατί για παράδειγμα τα τελωνία θα μπλοκάρουν τα εμπορεύματα. Για το Πακιστάν όπως έχετε καταλάβει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία ευθύνη αδειοδότησης. Ε, η απόφαση παροχής όπλων στην Ινδία και το Πακιστάν είναι απόφαση των εθνικών κυβερνήσεων, αν θέλουν ή όχι να παρέχουν όπλα στις χώρες αυτές. Ε, τώρα κοιτάξτε, εμείς τις συζητήσεις που έχουμε στην ΚΟΑΡΜ, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο η, το Ινδία και το, Ινδία και το Πακιστάν έχουν σοβαρούς λόγους αντιμετώπισης της πειρατείας, για παράδειγμα, στον Ινδικό ωκεανό, αλλά ε, και της τρομοκρατίας. Ε, υπάρχουν, για παράδειγμα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην περιοχή του Κασμίρου, που ε, ο κίνδυνος σύγκρουσης είναι πάρα πολύ μεγάλος. αυτά τα αγαθά συνήθως απορρίπτονται. Κάποια μπορεί να επιτρέπονται, γιατί υπάρχουν κάποιοι λόγοι ασφαλείας από πίσω, αλλά όμως όχι. Και αν δει κανείς τους, τον αριθμό των ε, απορρίψεων, μπορώ να σας πω ότι Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ε, συναλλαγών που δεν ε, γίνονται αποδεκτές για τους λόγους ευαισθησίας που αναφέρατε. Και όσον αφορά τώρα τα κριτήρια, κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις σε σχέση με την εφαρμογή των κριτηρίων Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην αξιολόγηση κινδύνου βάση των κριτηρίων και υπάρχει επίσης και η εθνική απόφαση που λαμβάνεται ε, ως ε, αποτέλεσμα αυτής της ε, αξιολόγησης κινδύνου βάσει των κριτήριων αυτών. Και αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο, το δέχομαι, βάσει της κανονικής δημοκρατικής ε, διαδικασίας. Δεν σημαίνει ότι τα κριτήρια είναι αμφισβητήσιμα ή δεν είναι καλώς διατυπωμένα, ε, αλλά αυτές οι αποφάσεις, αν είναι αμφισβητήσιμες, ε, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα κυρώσεις και όλα τελικά καταλήγουν στο ίδιο θέμα της, του δημοκρατικού ελέγχου επαφίεται στις πλέον, στους πλέον αρμόδιους δημοκρατικούς φορείς και στον ε, ε, εκτελεστικό ε, τομέα να κάνει ερωτήσεις και να ζητήσει κυρώσεις για την καλύτερη παρακολούθηση τώρα. Νομίζω ότι Υπάρχει ε, το θέμα της παρακολούθησης από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ξέρετε ότι υπάρχει παρακολούθηση των κυβερνήσεων ε, για τις εξαγωγές όπλων. Έχετε έναν αριθμό εθνικών κοινοβουλίων στο οποίο, στα οποία αυτό το θέμα συζητιέται πάρα πολύ έντονα ε, και άλλα κοινοβούλια στα οποία δεν αποτελεί ιδιαίτερο θέμα. Πάντως, ε, βάσει της ε, ε, μεγαλύτερης ευθύνης των εθνικών κυβερνήσεων, ξέρετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη παρακολούθηση και μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών. Ας σταματήσω εδώ καλύτερα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Lotton. Mr. Isbister. Κύριος ακούστηκαν πολλά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε ορισμένα. Αναφορά στον έλεγχο της τεχνολογίας έγινε από διάφορους ομιλητές και είναι ένας τομέας αυτός που είναι πάρα πολύ σημαντικός και από μια άποψη ενδεχομένως να είναι και πιο σημαντικός από την ε, κάθε αυτό εξαγωγή του εξοπλισμού διότι μπορεί να δώσεις με αυτόν τον τρόπο την τεχνογνωσία σε κάποιον να παράξει δικό του εξοπλισμό Άρα υπάρχουν διάφορες ε, επιπτώσεις. Και εγώ δεν βλέπω όσο θα ήθελα τουλάχιστον τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν ένα επιπλέον ε, επίπεδο ελέγχου. Ενώ σε κάθε μεγάλη συμφωνία υπάρχει, υπάρχουν διατάξεις και για την προστασία της εγχώριας παραγωγής. Το τι αποκαλύπτουν δηλαδή τα κράτη-μέλη προκειμένου να συνάψουν την εκάστοτε συμφωνία και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Διαφορετικά τα πράγματα στο πλαίσιο της συνθήκης για, την, ε, για το εμπόριο όπλων. Αυτό που έχω δει εγώ πολλές φορές είναι ότι κάθε συμφωνία που ε, περιλαμβάνει μεταφορά, τεχνο, ε, μεταφορά τεχνολογίας σε χώρα που έχει υπογράψει τη συνθήκη, θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνει ε, και ε, συζητήσεις για την προσχώρηση της εκάστοτε χώρας σε αυτήν την συνθήκη. Αν θέλεις δηλαδή να πάρεις αυτά τα όπλα πρέπει να υπογράψεις τη συνθήκη. Και βλέπω ότι δεν γίνονται αρκετά πράγματα. Όταν μιλώ σε αξιωματούχους για αυτό το θέμα, ε, μου λένε ότι δεν είναι πολύ ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση. Ενώ εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο πραγματικός ρεαλισμός. Τώρα, για τα όπλα που πουλήθηκαν στους ε, Σαουδάραβες, για τις βόμβες που χρησιμοποιούνται στα ε, μαχητικά αεροσκάφη που έχει εξαγάγει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Σαουδική Αραβία. Έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές στην Ιεμένη ή τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει σκοπός ε, να χρησιμοποιηθούν στην ΙΕΜΕΝΗ ε, ε, γιατί φαίνεται να έχει υπάρχει ξαφνικά μια αύξηση της ζήτησης και φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να δοθεί άδεια, να εγκριθεί η πώληση αυτή. Είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε. Υπήρξε αναφορά στο ζήτημα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Πολλά από τα επιχειρήματα που σχετίζονται με την απασχόληση και τις εξαγωγές όπλων βασίζονται σε μια αντίληψη ε, περί οικονομικών του 19ου αιώνα. Ότι αν ε, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα δεν υπάρχουν και θέσεις απασχόλησης. Είναι πολύ απλουστευτική αυτή η προσέγγιση. Ακριβώς διότι και το κεφάλαιο και η εργασία που έρχονται και συνεργάζονται στην βιομηχανία όπλων θα ε, προσπαθήσουν να, να κατευθυνθούν σε άλλους τομείς και σε άλλους κλάδους. Άρα ε, ενδεχομένως να υπάρχει και το, η περίπτωση να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης αν απελευθερωθούν ε, πόροι ε, και ανθρώπινοι που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην αμυντική βιομηχανία. Βεβαίως κάποιες πόλεις θα περάσουν δύσκολα. Αν ε, υπάρχουν εργοστάσια σε συγκεκριμένες πόλεις, προφανώς θα υπάρξουν προβλήματα στις πόλεις αυτές και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά παρόλα αυτά το επιχείρημα θα πρέπει να είναι κάπως πιο... Ε, εξελιγμένο από το να λέμε απλά ότι η αμυντική βιομηχανία δημιουργεί τόσες θέσεις απασχόλησης και αν την καταργήσουμε τότε θα χαθούν τόσες ε, θέσεις απασχόλησης. Για το κριτήριο 8, το κριτήριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει εδώ και χρόνια ε, νιώθουν μια απογοήτευση για το γεγονός ότι ε, αγνοείται το συγκεκριμένο κριτήριο από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν το λαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τους το συγκεκριμένο κριτήριο. Ε, θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ δύσκολη γιατί ε, ε, πολλές φορές ε, κατηγορούμαστε ότι είναι σαν να λένε οι πλούσιες χώρες τις φτωχές τι θα κάνουν και πώς θα αναπτυχθούν. Ένας νεοπικισμός δηλαδή ε, διακρίνεται πίσω από αυτό. Πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που το ζήτημα αφορά και την, ε, την ε, λελογισμένη ε, κατανομή των δαπανών. Άρα αν εξετάσουμε αυτό το, το έλογο έναντι του μη έλογου των δαπανών, ενδεχομένως να είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιληθεί αυτή αυτή αυτό το πρόβλημα. για την δεν εννοούσα πριν ότι είναι το ίδιο πράγμα οι εξαγωγέ όπλων στη Ρωσία και στην ε, ε, Ουκρανία. Απλά στην ε, περίπτωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία η Ουκρανία έθεσε το θέμα της κοινή θέση, ενώ στην περίπτωση των εξαγωγών όπλων προς την Ουκρανία το επιχείρημα αυτό το χρησιμοποίησε η Ρωσία. Δεν ήθελα να πω ότι είναι το ίδιο. Ήθελα ωστόσο να πω ότι θα πρέπει τα κριτήρια να ισχύσουν και όσον αφορά τις πωλήσει όπλων προς την Ουκρανία. Για την σύγκληση και την απόκληση. Να πω ένα θέμα που, ε, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πιάνο και την παρακολούθηση. Πολλές φορές ακούγεται το επιχείρημα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η παρακολούθηση ε, πρέπει να γίνεται από, την, από τη ΣΥΠΑ λόγω του ειδικού βάρους που έχουν. Ε, ενώ κανένα κράτο μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν, δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο όσον αφορά την παρακολούθηση της χρήσης των όπλων. Εγώ θα έλεγα ότι είναι Πράγματι, προβληματικό ε, η Τσεχία να λάβει μια τέτοια απόφαση, αλλά αν τα 28 κράτη-μέλη από κοινού αποφασίσουν ότι θέλουν να εφαρμόσουν μια κοινή πολιτική για την παρακολούθηση και να συνεργαστούν βεβαίως και στο πεδίο αυτό με τις ΗΠΑ, τότε ε, η προσέγγιση και η προοπτική αυτή είναι πολύ πιο ρεαλιστική. Και θα καλούσα τα κράτη-μέλη να το εξετάσουν το ενδεχόμενο αυτό σοβαρότατα. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να απάντησα. Thank you, Mr. Chair. όπως είπε και ο προλαλής σας, είναι δύσκολο να καλύψουμε τα πάντα, αλλά θα ήθελα να καλύψω ορισμένα πιο στρατηγική υφή ζητήματα από πλευράς βιομηχανίας. Ε, επειδή αναφέρθηκαν οι θέσεις απασχόλησης, θα ήθελα να σας πω ότι δεν μιλάμε για θέσεις απασχόλησης, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο στη βιομηχανία αυτή. Μιλάμε για 3.000 επιχειρήσεις και μιλάμε για ένα εκατομμύριο θέσεις. Το ίμιση αφορά την πολιτική αεροπορία και το άλλο μισό για τον τομέα άμυνας. Επίσης, αυτό που δεν έχουμε καλύψει στις 3.000 ε, επιχειρήσεις είναι οι 1.800 επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ε, έργο στον τομέα αυτό. Δηλαδή μιλάμε για πολλές θέσεις εργασίας. Ε, από πλευράς έρευνας και τεχνολογίας θα ήθελα να πω ότι υπάρχει η βάση για μια πολιτική άμυνας και ασφάλειας σε ευρωπαϊκό ε, ή εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν ε, και επιπτώσεις από τον τομέα ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία, στον τομέα της ιατρικής, ε, δορυφόρους και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε για εξαγωγές και όχι μόνο στη, για τη συνιστόσα ασφάλειας. Αλλά για να το κατανοήσουμε, θα ήθελα να πω ότι και από πλευράς βιομηχανίας δεν θα πρέπει να μιλάμε για το ευρωπαϊκό σκέλος ε, τεχνολογιών και άμυνας για την πρόθεση θέσεων εργασίας, αλλά για εξαγωγές. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Όταν μιλάμε για έλεγχο εξαγωγών, αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ένα μέρος μόνο του όλου πακέτου. Θα πρέπει να το θέσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιων προοπτικών, γιατί η κατάσταση δέκα χρόνια πριν ε, παρουσίαζε εντελώς διαφορετική εικόνα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λάβουμε αποφάσεις για το ε, μέλλον, όχι κάνοντας έναν προς τα πίσω αντικατοπτρισμό, αλλά ε, κάνοντας μια προβολή στο μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται περισσότερες δαπάνες ε, τα τελευταία χρόνια μέχρι το 2012 και εάν αποσύρετε τα αμερικανικά στοιχεία βλέπετε αύξηση και για το 2013-2014. Άρα ε, γίνονται μεγαλύτερες δαπάνες για τεχνολογίες άμυνας. Το 2013 και 2014 όλες οι περιοχές του κόσμου έκαναν περισσότερες αμυντικές δαπάνες η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να συρρυκνώσει τον προϋπολογισμό της. Αρχίσαμε με 400 δις και τώρα είμαστε σε 185 δις, δηλαδή έχουμε μια συρρήκνωση της τάξης του 60%. Αν δείτε πώς η Ευρώπη χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα που δαπανούμε, πόσα εντάσσονται στην ε, βιομηχανία, ε, είναι το 1 πέμπτον από τα 185 δις. Άρα μιλάμε για 35 δις. Ας το βάλουμε αυτό στο παγκόσμιο στερέωμα. Σήμερα δαπανούμε 15% της παγκόσμιας αγοράς. Και αν δείτε τι πάει πίσω στη βιομηχανία σε σχέση με τις ΗΠΑ, βλέπετε ότι το διπλό πάει πίσω στις ε, επιχειρήσεις σε σχέση με τις ΗΠΑ. Άρα, μιλάμε για ένα 8 με 10% της, ε, ε, των παγκοσμίων δαπανών και προσπαθούμε να προωθήσουμε έναν ηγετικό ρόλο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση. Ποιες είναι οι άλλες χώρες ε, και τι κάνουν ε, σε σχέση με την έρευνα και τεχνολογία. Το 2007 οι χώρες BRIC δαπάνησαν όσο η Ευρώπη όλοι μαζί. Το 2015 οι χώρες BRIC θα δαπανίσουν τρεις φορές ε, περισσότερο από την Ευρώπη σε σχέση με τις τεχνολογίες άμυνας. Άρα βλέπουμε μία μεταφορά οικονομικής και πολιτικής εξουσίας και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στις ε, τεχνολογικές ε, έρευνες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η εικόνα και αυτό σημαίνει πίεση και προς τις επιχειρήσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, πολλά διευθύνοντα στελέχη, πολλοί CEO λένε ότι θα πρέπει να ε, κινηθούν και σε επίπεδο μετόχων, γιατί πολλοί μέτοχοι λένε γιατί παραμένουμε σε αυτό το τομέα ε, τη στιγμή που υπάρχουν αναδυόμενες οικονομίες και αγορές. Μπορούμε να πάμε σε εκείνες, δηλαδή στο κάτω μέρος της ε, αλυσίδας ε, προμηθείων. Αλλά εάν δεν προωθήσουμε την έρευνα και τις τεχνολογίες, πώς θα κρατήσουμε τη θέση μας σε αυτή την αλυσίδα αξιών. Γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε ανταγωνιστικά από πλευράς ε, Ευρώπης. Θα πρέπει να κινηθούμε ανάντι, γιατί πολλοί νέοι ε, μηχανικοί θέλουν να μπουν σε αυτό το τομέα και λένε γιατί να ε, μπω σε αυτό τον τομέα και να μην πω στην πολιτική αεροπορία που έχει μέλλον για τους ε, νέους μηχανικούς. Ε, εάν συζητήσουμε την ευρύτερη εικόνα, οι εξαγωγές είναι το σημαντικότερο κομβικό στοιχείο. Μιλάμε για στρατηγική αυτονομία, πώς θέλουμε να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας για να επικρατήσουν και τι σημαίνει αυτό ως προς τις τεχνολογικές και στρατιωτικές μας ικανότητες, πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την αλυσίδα, την προμηθευτική αλυσίδα και υπ' αυτή την έννοια οι εξαγωγές είναι ένα μέσον για να προωθήσουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τις άμεσες, αμεσότερες ερωτήσεις, κατά πόσο η Ευρώπη είναι πραγματικά ανταγωνιστική σήμερα, πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και στην Ευρώπη για να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα έχουμε να κάνουμε με μια κατακαιρματισμένη κατάσταση και η βιομηχανία εδώ και πολύ χρονικό διάστημα μιλά για την εναρμόνιση στρατιωτικών απαιτήσεων, αν και είμαστε 28 δεν θα πρέπει να παρά να εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας, δηλαδή να γίνονται μεγαλύτερες προμήθειες από περισσότερα κράτη-μέλη από κοινού. Αυτό θα το καλωσόριζε η βιομηχανία. Υπάρχουν νικητές και ιτημένοι, αλλά η βιομηχανία θέλει να γίνει αυτή η συζήτηση και προώθηση και είναι κάτι που θα οδηγούσε σε μια αναπτυξιακή ε, διαδικασία γιατί οι συγχωνεύσεις σχετίζονται με την αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών για την βελτιστοποίηση των ε, προσπαθειών. Μιλάμε για την διαδικασία επιμερισμού, ε, σύγκλησης, pooling. Θα πρέπει να δούμε τι σκέφτονται οι αρχές στα διάφορα, στα διάφορα κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα που εφήγει είναι κατά πόσο εστιάζουμε την προσοχή μας στους βραχυπρόθεσμους στόχους ως προς εξαγωγές. Ναι, ίσως να γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί αν δείτε τι κάνει η βιομηχανία αυτή έπρεπε να επαναπροσανατολίσουμε τις εξαγωγές μας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δούμε πού θα βρούμε τις αγορές, πού υπάρχουν οι πελάτες, πού υπάρχουν ανάγκες. Εκεί θα πρέπει να κινηθείτε και να δείτε κατά πόσο αυτό συμβαδίζει με την εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων. Υπάρχουν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να χρειαστεί και πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι που αλλάζει εν μία νυχτή, αλλά όταν κινούμαστε προς την παγκόσμια αγορά θα πρέπει να κινηθούμε προς τους πελάτες. Και επειδή δεν υπάρχει στρατηγικός διάλογος για την ευρωπαϊκή αυτονόμηση, Μιλάμε για την επιβίωση της βιομηχανίας και ίσως αυτό να μην ήταν και το πιο ρεαλιστικό μέχρι τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να πω ότι έγινα λόγος και για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Όπως σας είπα, αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί και η Transparency International, ο οργανισμός αυτός, έχει ένα δίκτυο κατά της διαφθοράς. Και ε, αυτό αφορά όχι μόνο τη βιομηχανία, αλλά και τα κράτη, γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και από πλευράς καταναλωτών. Όταν υπάρχει διαφθορά δεν υπάρχουν παραχαμένοι και αυτό τον γνωρίζουν οι, όλες οι βιομηχανίες ε, έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μικρότερες δεν ενδιαφέρονται, αλλά δεν έχουν την πυγμή να μπουν στην αγορά. αλλά η βιομηχανία έχει την δική της ε, διαδικασία. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η η διαδικασία αδειοδότησης, αλλά όλες αυτές οι παράμετροι. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο ε, μέσα στα πλαίσια της αδειοδότησης ζητείται άδεια από μια συγκεκριμένη ε, κυβέρνηση και πολλές φορές δεν υπάρχει έγκριση από την ε, κυβέρνηση γιατί λέει η κυβέρνηση «Α, είναι πολύ, ε, πολύ επικίνδυνο γιατί αυτή η χώρα έχει υψηλή διαφθορά, άρα δεν θα το κάνουμε». και θα πρέπει να συγκρίνουμε τι κάνει η ε, Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ. Αν δείτε το επίπεδο φιλοδοξίας τον είπα, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μία μεταφορά στο οικονομικό και πολιτικό σκέλος και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδώσουμε μια κατάσταση παγκόσμιας ασφάλειας. Μιλάμε για τεχνολογίες τα τελευταία. Μιλάμε για στρατιωτικές ικανότητες, για κέπα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς προωθούμε τις τεχνολογίες μας και πώς είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει η ικανότητα για να υποστηρίξουμε το επίπεδο φιλοδοξιών μας. Άρα θα θέλαν να προωθηθεί η νέα γενναιά τεχνολογία της ΕΠΑ μέσα στα πλαίσια αυτών των ικανοτήτων χωρίς να ε, είμαστε, είμαστε σίγουροι ποια είναι τα σημεία ζωτικής σημασίας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς να κινηθούμε στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές μας ε, επιδιώξεις. Κάτι το, στο οποίο υπολοιπόμεθα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μία, ε, μία ερώτηση πληρωματική ε, στον κύριο Πίο που δεν έχει να κάνει άμεσα με τον έλεγχο των εξαγωγών Η Ελλάδα είναι μάλλον ε, ήταν αρκετά ε, μεγάλος αγοραστής ε, όπλων και εντός της Ένωσης αλλά και εκτός παρά την τεράστια κρίση. Ποια είναι η άποψη του κλάδου προς αυτό Φαντάζομαι ότι δεν ήταν εμπορικά τα δάνεια, ήταν ε, μέσω των τραπεζών. Αλλά ποια είναι η άποψη του κλάδου σε σχέση με την ε, κατάσταση της Ελλάδας. Υπάρχουν ε, κάποιοι λόγοι που αφορούν για παράδειγμα το χρέος. Αυτό που έχουμε δει ως τώρα ε, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτε την ερώ... για το συζήτηση ε, για την Ελλάδα, κατά πόσο η Ελλάδα δηλαδή είναι καλύτερος ή λιγότερο καλός πελάτης από άλλου. Εγώ δεν βλέπω καμία τέτοια συζήτηση, ούτε καν στο υψηλότερο επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, έτσι ολοκληρώνεται η πρωινή μας συνεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, τρεις προσκεκλημένους μας για την ε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και περιεκτική παρουσίασή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και παρακαλώ πολύ ε, να παραστείτε σήμερα το απόγευμα στην κοινή μας συνεδρίαση για τις ε, παγωμένες συγκρούσεις και την κατάσταση ασφαλείας ε, στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ.